c'est toujours le, le compromis sans la mienne, de compromis sans. Bueno, eh, buenos días a... Καλή σας μέρα. Ξεκινάμε τις συνεδρίες της Επιτροπής Αλίας. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, την εγκρίνουμε. Δεύτερον, Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίας, το, της συνεδρίας της 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2009. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα τα θεωρήσουμε ως εγκεκριμένα. Τέταρτον. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Την περασμένη εβδομάδα παρέστημε στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας στην, ε, της Αντιπροσωπείας Αλίας στην χώρα των Βάσκων συνεδρία ήταν πολύ καλή, πολύ ωφέλιμη και ενδιαφέρουσα για όλους όσους παρέστημεν στην ε, αυτόν την περιοχή της χώρας των Βασκών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μπιλμπάου που είχε αναλάβει την οργάνωση. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Την ευχαριστώ παρόλα αυτά. Σημείο 5 της ημερησίας διάταξης. Έκθεση σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής. Έχουμε κατάλογο ψηφοφορίας. Προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης. Συγητής ο κύριος Αρσένης. Το θέμα έχει συζητηθεί. 4 Φεβρουαρίου ήταν η ημερομηνία για πολυτροπολογιών. τροπολογιών. 35 υποβλήθηκαν. Ο κύριος Αρσένης δεν ξέρω αν θέλει το λόγο, αλλιώς να περάσουν στην πληροφορία. Thank you very much. Ε, Λάβαμε όλες τις ε, τροπολογίες και έχουμε υποβάλει και προτάσεις συμβιβασμού. Ε, συζήτησαμε και με τον κύριο Χάντεκ και με άλλους συναδέλφους. Νομίζω με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συμπεριλάβουμε τις απόψεις όλων των συναδέλφων. Ελπίζω το αποτέλεσμα να ικανοποιήσει τους πάντες. Ε, Ευχαριστώ. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας. Περνάμε στην ψηφοφορία. Καταρχήν, συμβασμός υπαριθμών 1 για την παράφο 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Ξανα... Α, ξαναρχίζουμε. Ξαναρχίζουμε. Άρχεται η ισοφορία. Υπάρχουν άλλα προβλήματα ή εντάξει όλοι. A ver, αλλάξτε θέσεις αν θέλετε, να δείτε πώς λειτουργούν οι διπλανές κονσόλες. Βάλτε τους στο on. Άρχεται η ψηφοφορία. Εντάξει, ωραία. Εντάξει, κλείει η ψηφοφορία. Se cierra la votación. 11 eh, υπέρ. Εγκρίνεται. Καταπίτη τροπολογία 1, 2, 4. Οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία της κυρίας Πατράου Νέβες, την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. 7 υπέρ. Κυρία Λεβά, το ίδιο πάλι. Δεν ψήφισα. Δεν πρόλαβα να ψηφίσω. Κλείσα την ψηφοφορία πολύ γρήγορα. Να ξαναψηφίσουμε αργά-αργά. Ναι. Άρχεται η ψηφοφορία της τροπολογίας 3. Ωραία. Κλείνουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Οκτώ ψήφοι υπέρ. Ψηφίζουμε την τροπολογία πέντε. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τον δεύτερο, τη δεύτερη συνεργαστική πρόταση. Άρχεται. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 6, 7 και 8. Ψηφίζουμε την τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 10. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Περνάμε στο συμβαστική πρόταση παριθμών 3. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 14, 13, 11, και 12. Ψηφίζουμε την 16. Άρχεται. Λίγη. Ε, Απορρίπτεται. Τροπολογία παριθμό 15. Άρχεται. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 8 υπέρ 6 κατά. Συμβιβασμό υπαριθμών 4. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 17 και 18. Συμβαστική πρόταση υπαριθμών 5. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι τροπολογίες 21, 22, 23 και 24. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 25. Μια προστίκη. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση υπαριθμών 6. Άρχεται. Δεν Εγκρίνεται. Καταπίπτουν οι 19, οι 20, 27, 28, 29, 30 και 32. Ψηφίζουμε την συμβαστική πρόταση παριθμών 7. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Καταπίπτει υπαριθμών 33. Ψηφίζουμε τη συμβαστική πρόταση υπαριθμών 8. Άρχεται. Λίγη. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η 26 και η 35. Ψηφίζουμε την τροπολογία υπαριθμών 34. Άρχεται. Λίγη. 8 υπέρ 7 κατά. Εγκρίνεται λοιπόν. Ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση στο σύνολό τη όπω τροποποιήθηκε. Άρχεται. Λίγη ψηφοφορία. Συγχαρητήρια κύριε Αρσένη. Ομοφωνία. 15 ψήφοι υπέρ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ανταλλαγή απόψεων με την νομική υπηρεσία του, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την νομική γνωμοδότηση της 13ης Ιουλίου 2009 για τη Συμφωνία Σύμπραξης με το Μαρόκο. Η γνωμοδότηση αυτή ζητήθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξη την περασμένη θητεία με πρόεδρο τον κ. Μπορέλ Η ομάδα των Πρασίνων ζήτησε το ζήτημα να συζητηθεί και στη δική μας Επιτροπή. Στην προηγούμενη συνεδρίασή μας είχε προβληθεί στην ημερήσια διάταξη. Ο τύπος ε, με συκοφάντησε ότι εγώ σαμποτάρισα τη συζήτηση και δεν συζητήθηκε. Όχι, απλά δεν είχαμε χρόνο, εσείς το ξέρετε. Τη βάλαμε, το βάλαμε λοιπόν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Δεν ξέρω ποιος μίλησε για σαμποτάζ στον τύπο. Ε, ήταν άδικη, αυ, άδικος αυτός ο χαρακτηρισμός. Θα δώσω το λόγο στον, τον κύριο Πάσος να μας παρουσιάσει την ομοδότηση. Να κάνω μια παρουσίαση 15 λεπτών, αν μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε. 15 λεπτά είναι εντάξει. Όσο χρειάζεστε. Δεν θέλω να με κατηγορήσουν ξανά για σαμποτέρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περίπλοκο νομικό θέμα. Η ελευτική συμφωνία με το Μαρόκο. Έχουμε δύο επιτροπές στο Κοινοβούλιο που έχουν δραστηριοποιηθεί στο ΜΕΑ, Επιτροπή Ανάπτυξης και η δική σας. Και η νομική υπηρεσία γνωμοδότησε δύο φορές Καταρχάς, όταν επρόκειτο να συναυθεί η συμφωνία, τέλος διαπραγματεύσεων, Ιανουάριο 2006, και το ερώτημα που είχε τεθεί τότε στην νομική υπηρεσία ήταν κατά πόσο ο κανονισμός του Συμβουλίου για τη Σύνοψη Συμφωνίας με το Μαρόκο θα επέτρεπε σε σκάφη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να αλλιεύουν στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας και αν αυτό ήταν συμβατό με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και ετοιμάσαμε άλλη νομική γνωμοδότηση το Μάιο του 2009 που έχει διαβιβαστεί στα μέλη που ζητήθηκε από τον κύριο Μπορέλ όπως είπατε και το ερώτημα ήταν το εξής εφόσον η πρώτη νομική γνωμοδότηση του 2006 εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να λιεύουν τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ενώσεω στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας μετά από δυόμιση χρόνια, όταν υπευλήθη το Μάιο του 2009 η αίτηση, ήταν σαφέ ότι τα σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω αλίευαν στα ύδατα τη Δυτική Σαχάρα. Άρα το ερώτημα του κυρίου Μπορέλ ήταν κατά πόσο, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στοιχεία περί αλλιευμάτων των σκαφών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που αλίευαν στα ύδατα τη Δυτική Σαχάρα, κατά πόσο αυτό ήταν σύμφωνα με τι αρχέ του διεθνού δικαίου. Οι δύο νομικέ γνωμοδοτήσει είναι αλληλένδετε. Μία δόθηκε πριν από την Σύνευση συμφωνίας του 2006 και άλλη το 2009. Μετά από τριετία της ε, υλοποίησης της συμφωνίας. Αν με επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, θα κάνω την παρουσία μου σε τρία τμήματα. Το πρώτο τμήμα αφορά την κατάσταση όσον αφορά το διεθνές δίκαιο στη Δυτική Σαχάρα και ποιες είναι οι ευθύνες του Μαρόκου. Δεύτερο τμήμα, κατά πόσο είναι συμβατό αυτό η Συμβατή Συμφωνία του Διεθνές Δίκαιο όταν συνήφθη το 2006 και το τρίτο τμήμα, το σημαντικότερο για σας, αφορά τη συμβατότητα της Συμφωνίας του Διεθνές Δίκαιο σήμερα ως υλοποιείται μέχρι τούδε. Το πρώτο τμήμα, η κατάσταση, ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά το διεθνές δίκαιο της Δυτικής Σαχάρας και ποιο είναι το νομικό καθεστώς της διεθνου, στο διεθνές δίκαιο της Δυτικής Σαχάρας. Είναι γνωστό ότι η Δυτική Σαχάρα είναι μια, ένα έδαφος, μια επικράτεια που δεν αυτοδικείται εν τη ενία του άρθρου 73 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Βεβαίως είναι παλιά ιστορία η ιστορία της Δυτικής Σαχάρας. Δεν μπορώ να επισέθω σε λεπτομέρειες, όμως αρκεί να πούμε ότι η Δυτική Σαχάρα ήταν ισπανική απικία το 1884 και παρέμεινε υπό Ισπανική κυριαρχία μέχρι ότου αποχώρησε το 1976 η Ισπανία. Κατά τη διάρκεια της Ισπανικής διοικήσεως, η Δυτική Σαχάρα συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των μη αυτοκυβερνούμενων περιοχών και ακολουθούσε το άρθρο 73 της χάρτας του ΙΕ Ισπανία. Σημαντικό να σας πω τι λέει το άρθρο 73. Το άρθρο αυτό λέει ότι τα μέλη του ΟΗΕ που έχουν υπομειστεί ευθύνες για τη δίκηση εδαφών των οποίων οι λαοί δεν έχουν πλήρη αυτοδιοίκηση, αυτοδιάθεση, αναγνωρίζουν την αρχή σύμφωνα την οποία τα συμφέροντα των κατοίκων αυτών των εδαφών είναι πρωτής σημασία και δέχονται σαν ιερό, ιερή την υποχρέωση να σέβονται ε, το, τη διαβίωση, το επίπεδο διαβίωση των κατοίκων της περιοχής. Όταν αποχώρησε η Ισπανία το 1976, το Μαρόκο και η Μαυριτανία κατέκτησαν την περιοχή παρά την αντίσταση του κινήματος Πολυσάριο. Και το 1976 το κίνημα αυτό ανακοίνωσε την εξαρτησία του, προκήρυξε την εξαρτησία του, δεν αναγνωρίστηκε η ανεξαρτησία από πολλά κράτη το ΙΕ και το 1976 το Μαρόκο και η Μαυριτανία διέρεσαν την ε, κράτη Δύο τρίτα για το Μαρόκο, ένα τρίτο για τη Μαυριτανία. Το 1979 η Μαυριτανία αποχώρησε και αναγνώρισε την ε, Αραβική Δημοκρατία τη Σαχάρα και το Μαρόκο ε, κατέξε αυτή την περιοχή και ύποψε τείχος ύψος 3 μέτρων, μήκους 2.000 χιλιόμετρων και απέκοψε τη δική Σαχάρα. Το 1988 το Μαρόκο και το Πολυσάριο ε, υπέγραψαν μια συμφωνία διευθέτησης που προωθήθηκε από τον ΙΕ και από την ε, οργάνωση των αραβικών χωρών μέσω για τη διοργάνωση ενός δημοσιοφίσματος. Και ποιο ήταν το σχέδιο. Το σχέδιο μάλλον υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας το 1990. Κοίτα the Secretary General of the United Nations appointed a special representative and a UN mission, the MINURSO, has been created. The difficulty for the organisation of the referendum was the identification of those entitled to vote. Δεν μπορούσαν να εντοπιστούν εκείνοι που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν. Και το Μαρόκο ήθελε να συμπεριλάβει πολλούς επίκους που είχαν μετακινηθεί από το Μαρόκο που άλλαξε τη δημογραφική σύνδεση της περιοχής και υπήρξαν προβλήματα που σχετιζόταν με πολλούς πρόσφυγες από τη Σαχάρα που ζούσαν σε άλλες χώρες. Ένα άλλο πρόβλημα ήταν ποιο πεδίο κάλυπτε το δημοψήφισμα, αυτονομία ή ανεξαρτησία και πώς θα μπορούσε να εφαρμόσει κανείς το ενδεχόμενο αποτέλεσμα, αν το αποτέλεσμα ήταν ανεξαρτησία. Τούτων λεχθέντων, κυρία Πρόεδρε, το νομικό καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας είναι ότι είναι ε, δεν έχει αυτοδιάθεση η περιοχή, όπως λέει το άρθρο 73 της Χάρτας των Ηνωμένων Θεών. De facto ελέγχει το Μαρόκο το μεγαλύτερο τμήμα των εδαφών. Δεν αλλάζει το καθεστώς της περιοχής ότι είναι μη αυτοδιοικούμενη περιοχή. Ποιες είναι οι συνέπειες σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Εγώ βλέπω τέσσερις συνέπειες. Η πρώτη είναι ότι το άρθρο 73 της χάρτας ισχύει. Το δεύτερο είναι ότι το Μαρόκο δεν είναι διοικητική εξουσία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, αλλά de facto κυβέρνηση της Δυτικής Σαχάρας. Τρίτον, ακόμα και αν το Μαρόκο δεν έχει το καθεστώς δύναμης κυβερνητικής, η Δυτική Σαχάρα είναι μη αυτοδικούμενη περιοχή. Και αυτό σημαίνει ότι η εκμετάλλευση πόρων στη Δυτική Σαχάρα δεν είναι κάτι παράνομο αυτό καθεαυτό, εκτός αν αγνοούνται οι ανάγκες, τα συμφέροντα και τα ωφέλη των λαών της περιοχής όταν γίνεται εκμετάλλευση αυτών των πρώτων Ήδη κατά το παρελθόν συνήθισαν δύο συμβάσεις του Μαρόκου με ξένες εταιρείες όταν ετέθη το θέμα τη συμβατότητα αυτή τη προσέγγιση με το διεθνέ δίκαιο. Και ο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ διόρισε τον κύριο Κορέλ που είναι υπεύθυνο για τα νομικά θέματα, το ΙΕ, που κατέληξε σε νομική τοποθέτηση και είπε σαφώ ότι αυτέ οι συγκεκριμένε συμβάσει, αυτέ καθεαυτέ δεν ήταν παράνομε, διότι είναι συνεπάγονται εκμετάλλευση ό,τι φυσική αφαίρεση των φυσικών πόρων, όμω εάν περαιτέρω εξερεύνηση, ανείχνευση και εκμετάλλευση ε, και δραστηριότητε εκμετάλλευσεως γινόταν χωρί να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των λαών τη Δυτική Σαχάρα, τότε θα παραβιαζόταν οι αρχέ του Διεθνού δικαίου που αφορούν του ορυκτού πόρους και τι συναφεί δραστηριότητε σε μη αυτοδικούμενε περιοχέ. Λοιπόν, βασική όρη στη νομική γνωμοδότηση ποιοι είναι, ότι τα συμφέροντα και επιθυμίε των λαών της Δυτικής που να λαμβάνονται υπόψη πώς να εφαρμόζονται αυτές οι αρχές τώρα στο τι γίνεται σήμερα και στην περίπτωση της αλληλευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο. Αυτό αφορά το δεύτερο κομμάτι της παρουσιάσής μου. Ήταν η κατάσταση όταν συνήθη η συμφωνία και ποια είναι η σημερινή κατάσταση. Όταν συνήθη η συμφωνία εκπονήσαμε την πρώτη νομική μας γνωμοδότηση. Όταν συνήθη συμφωνία δεν ήταν σαφές κατά πόσο εκάλυπτε τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Όμως το παράρτημα 2 του πρωτοκόλου ανέφερε ότι για βιομηχανικό πε, ε, πελαγική ε, εκμετάλλευση ε, βόρεια του 29ου ε, παραλίλου ε, μπορούσε να γίνει νότια του 29ου παραλίλου καλυπτόταν τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Υπόθηκε λοιπόν ότι οι αλληλευτικές συμφωνίες, η αλληλευτική συμφωνία που συνήφθη δεν ήταν παράνομη αυτή καθεαυτή, ανάλογα το πώς εφάρμοζε τη συμφωνία το Μαρόκο και για να την εφαρμόσει τη συμφωνία το Μαρόκο θα έπρεπε να λάβει υπόψη τα συμφέροντα των τόπιων πληθυσμών της Δυτικής Σαχάρας. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα μετά από μια τριετία της εφαρμογής της συμφωνίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία σήμερα τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πηγαίνουν εκεί και αλλιεύουν στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το είπε επανειλημμένα, αυτό είναι σίγουρο και αρκετά ερωτήματα ετέθησαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού και μία είχε τεθεί προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν η κυρία Φρίντα Μπρέπελς το ερώτημα τον Αύγουστο ετέθη του 2008 και ρωτά πώς αυτή η συμφωνία ωφελεί τους ντόπιου πληθυσμούς της Δυτικής Σαχάρας και απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 12 Σεπτεμβρίου του 2008 και είπε «Γαλλιστή, σύμφωνα με ερμηνεία του Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ, το Μαρόκο, παρόλο που δεν αναγνωρίζεται από τον ΙΕ ως δεζούρι διοικητική αρχή, μπορεί παρόλα αυτά να συνά τις συμφωνίες όσον αφορά τους φυσικούς πόρους της Δυτικής Σαχάρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ντόπιοι πληθυσμοί μπορούν να ωφελούνται από αυτές τις συμφωνίες. Θεωρούμε λοιπόν ότι εναπόκειται στο Μαρόκο να λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίζει την εφαρμογή της συμφωνίας σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του διεθνούς δικαίου. Και προσθέτει όσον αφορά τα ωφέλη για τον πληθυσμό, για τους πληθυσμούς της Δυτικής Σαχάρας, η τομεακή πολιτική της αλίας του Μαρόκου που υποστηρίζεται από την Συμφωνία Εταιρική Συνεργασία στην Αλία θα πρέπει να υποστηρίξει την ανάπτυξη του τομέα στη Δυτική Σαχάρα που άμεσα θα ωφελεί τους τοπικούς πληθυσμούς και του προσελήφθησαν ναύτες από την περιοχή από τους πλειοκτήτες των σκαφών της ευρωπαϊκή Ενώσεως που αλλιεύουν στη Δυτική Σαχάρα και ιδιωτικέ επενδύσεις ευρωπαϊκές που συνδέονται άμεσα με την εφαρμογή της συμφωνίας έχουν δρομολογηθεί και δημιουργούν προστιθέμενη αξία και νέες θέσεις ε, εργασίας. Οπότε είναι ξεκάθαρο τώρα ότι μπορούμε να πούμε ότι τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πηγαίνουν εκεί και ότι εφαρμόστε και συμφωνία προς όφελος και κέρδος των λαών της ε, Σαχάρας. Όμως το πρόβλημα είναι κατά πόσο έχουμε επαρκείς πληροφορίες. Το ερώτημα είναι, έχουμε αρκετές πληροφορίες που να μας οδηγούν στο να πιστεύουμε ότι η συμφωνία εφαρμόζεται με έναν τρόπο που ωφελεί τους λαούς της Δυτικής Σαχάρας. Και εδώ η απάντηση δεν είναι καταφατική. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες στον αφορά το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε αυτή την απάντηση το Σεπτέμβριο του 2008. Η Μικτή Επιτροπή συνεδριάζει μία φορά το χρόνο. Συνεδρίασε την προηγούμενη φορά 2 και 3 Φεβρουαρίου ενεστώτος έτους και η κατάσταση παραμένει ασαφής κατά τη δική μας άποψη. Νομικός, ο σεβασμός των διεθνών νόμων για την εφαρμογή της Ελευτικής Συμφωνίας είναι κάτι που δημιουργεί πρόβλημα. Είναι προφανές ότι η Ένωση υποχρεούται να σεβαστεί τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και αληθεύει ότι η συγκεκριμένη κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα είναι πραγματικά περίπλοκη. Το δημοψήφισμα ποτέ δεν διοργανώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη και τα Ηνωμένα Έθνη σίγουρα πρέπει να βρουν μια λύση. Όμως, παρόλο και είναι περίπλοκη η κατάσταση, και είναι περίπλοκη η αξιολόγηση του κατά πόσο η συμφωνία λευτική ωφελεί τους λαούς της Σαχάρας, το πρόβλημα οφείλεται γιατί είναι και ένα απόσπαστο τμήμα του Μαρόκου για το Μαρόκο και για το Εμπολισάριο αυτό τα εδάφη δεν ανήκουν στο Μαρόκο. Εν τω μεταξύ βλέπουμε τρεις λύσεις για το πρόβλημα κυρία Πρόεδρε. Βεβαίως από νομική σκοπιά θα τα αναφέρω. Η νομική υπηρεσία δεν θα σας πει πολιτικός πώς ποια είναι η καλύτερη λύση. Εγώ βλέπω τρεις δυνατότητες νομικής φύσεως λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα του μη σεβασμού των διεθνών νομικών υποχρεώσεων. Μία δυνατότητα λοιπόν που υπάρχει. Να εφαρμοστεί η συμφωνία με έναν τρόπο με τον οποίο εξαιρούνται τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υποβάλει, δεν θα δώσει άδειε αλίας που θα φορούν αλία στα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας. Αυτό βεβαίως, ακόμα και αν είναι νομικά εφικτό, δημιουργεί πρόβλημα οικονομικού ρεαλισμού, διότι καταβάλλονται χρήματα, γίνονται πληρωμές για αλεία σε αυτά τα ύδατα. Άλλη δυνατότητα, η δεύτερη. Αναστολή της συμφωνίας. Άρθρο 15 της συμφωνίας αναφέρει ότι η εφαρμογή της εν λόγω συμφωνίας μπορεί να ανασταλεί κατόπιν πρωτοβουλίας ενός των συμβαλωμένων μερών σε περίπτωση σοβαρής διαφωνίας όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Αυτή είναι μια δεύτερη δυνατότητα. Η τρίτη δυνατότητα είναι η εξή. Και είναι και πιο ρεαλιστική ενδεχομένω. Η συμφωνία να φεθεί να ακολουθήσει την πορεία της μέχρι ότου να εκπνεύσει. Διότι η συμφωνία είναι τετραετής. Ξεκίνησε 28 Φεβρουαρίου του 2007 και θα εκπνεύσει 28 Φεβρουαρίου 2011 σύμφωνα με το άρθρο 12 της συμφωνίας. Η συμφωνία, και αυτό είναι σημαντικό που λέω, η συμφωνία θα, ανανεωθεί, θα ανανεώνεται ανά τετραετία, εκτός εάν ανακοινωθεί ο τερματισμός αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 14. Το άρθρο 14 αναφέρει το μέρος που θέλει να τερματιστεί η συμφωνία θα πρέπει να κοινοποιήσει γραπτό στην πρόθεσή του να αποσυρθεί τουλάχιστον ένα εξάμεινο πριν την εκπνοή της συμφωνίας. Αν το Κοινοβούλιο λοιπόν και η Επιτροπή σας πιστεύει ότι υπάρχει πρόβλημα, αν δεν πούμε τίποτα, η συμφωνία αυτομάτως σιωπηρά ανανεώνεται για άλλη μια τετραετία. Αν όμως θέλουμε αυτή η συμφωνία να σταματήσει όταν εκπνεύσει στην τετραετία, δηλαδή 28 Φεβρουαρίου του 2011, τότε θα πρέπει να αντιδράσουμε γραπτός πριν τις 28 Αυγούστου φέτος. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω τυχόν ερωτήσεις σας. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Φοντάνα. Ε, η κυρία Φοντάνα, ο κ. Φοντάνα. Ευχαριστώ για αυτή την νομική γνωμοδότηση των υπηρεσιών του Κοινοβουλίου να πω λίγα πράγματα χωρίς να μπω σε κάποια νομική συζήτηση κάποιο διάλογο με την νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με την νομική υπηρεσία της Κομισιόν, να σας πω ότι αυτή η συμφωνία είναι συμβατή με το Διεθνές Δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της στο πλαίσιο της τελευταίας μικτής επιτροπής που έλαβε χώρα στις 2 και 3 Φεβρουαρίου, τα θέματα αυτά συζητήθηκαν Η επιπτώσει τη συμφωνία σε ό,τι αφορά τι ε, αλευτικέ δραστηριότητε και την υποστήριξη του τομέα και η Κομισιόν βρίσκεται σε μόνιμο διάλογο με το Μαρόκο για αυτό το θέμα. Επιβλέπει την εφαρμογή της συμφωνίας και δεν διαθέτουμε καμία πληροφορία που να μας πείθει ότι οι αλευτικές δραστηριότητε που λαμβάνουν χώρα δυνάμει της συμφωνίας δεν είναι υποφελείς για την Δυτική Σαχάρα. Ευχαριστώ κύριε Φοντάνα. Κύριο Ζωμέβα. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ικανοποιημένο που έχουμε αυτή την ευκαιρία για τη σημερινή συζήτηση. Γιατί έχουμε, έχει περάσει πολύ καιρό που περιμένουμε. Πρέπει να πω ότι δεν βρήκαμε Τίποτα καινούριο. Το πρόβλημα, αν το έχω καταλάβει καλά, είναι ότι είναι αλήθεια ότι μπορεί η συμφωνία να είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο, όπως λέει Κομισιόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόζεται και σωστά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αν η θέση μας είναι ότι δεν έχουμε επαρκείς πληροφορίες ότι η εφαρμογή της συμφωνίας είναι ωφέλιμη για τους πληθυσμούς της Σαχάρα, ίσως να μην έχουμε ρωτήσει τους σωστούς ανθρώπους. Γι' αυτό συμβαίνει αυτό. Προφανώ, αν μιλούμε μόνο με τι αρχέ του Μαρόκου, δεν θα μα πούν ότι είναι επιζήμιο για του πληθυσμού τη Σαχάρα η συμφωνία. Έχουμε και πολλέ πληροφορίε από από ανθρώπου που προέρχονται ακριβώ από τα μέρη που υποτίθεται ότι ωφελούνται από αυτή τη συμφωνία και έχουν τελείω διαφορετική άποψη για την κατάσταση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν εμεί ψηφίσαμε τη συμφωνία το 2006, πολλοί καταψήφισαν στο Κοινοβούλιο γιατί δεν ήταν απόλυτα σαφέ ποιο ήταν το εύρο του πεδίου εφαρμογή. Τώρα επιβεβαιώθηκε ότι αυτό ίσω να είναι ένα από τα προβλήματα. Γιατί μπορεί να είναι σωστό να συμπεριλάβουμε τα ύδατα της Δυτικής Σαχάρας εάν αυτό είναι ωφέλιμο για τους πληθυσμούς της περιοχής αλλά εξακολουθεί να ισχύει ότι εξακολουθεί να είναι δυνατότητα να παραμείνουν εκτός της συμφωνίας τα ύδατα της Σαχάρας. Ίσως να μην είναι πολύ ρεαλιστικό, αλλά παραμένει μία πιθανότητα. Οπότε, ερώτημα προς την Κομισιόν. Εφόσον δεν έχουμε σχετικές ή σαφείς πληροφορίες για την εφαρμογή της συμφωνίας, ότι δηλαδή είναι ωφέλιμη για τους πληθυσμούς της Δυτικής Σαχάρας, εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον πρέπει να ανασταλεί. Τουλάχιστον να ανασταλεί, αν μη τι άλλο, η συμφωνία. Οπότε εδώ μπορούμε να το δούμε και από την αντίθετη πλευρά. Ας μην περιμένουμε μέχρι να βρεθούν ε, αποδείξεις για να ακυρωθεί η συμφωνία. Η απόδειξη πρέπει να είναι για να συνεχιστεί η συμφωνία ότι όντως είναι θετική και είναι επωφελής για τους πληθυσμούς. Και αν αυτό μπορούμε να το πετύχουμε και σε πολιτικό και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε νομικό, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Γιατί και εμείς εποφελούμεθα από αυτή την εκμετάλλευση. Κάποια, ε, ε από το, κάποια σκάφη από το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν εποφεληθεί. Επομένως είναι και δική μας ευθύνη να εγγυηθούμε ότι η εκμετάλλευση αυτών των υδάτων είναι προς όφελος του πληθυσμού της Δυτικής Σαχάρας. Οπότε υπάρχει διπλή ε, ευθύνη και από τη δική μας πλευρά και από την άλλη πλευρά. Δεν βλέπω άλλη λύση εγώ προς το παρόν, παρά μόνο να αναστείλουμε τη συμφωνία. Δεν έχουμε λόγο να συνεχίζουμε την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας υπό αυτέ τι συνθήκε τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την νομική υπηρεσία που μας έκανε την παρουσίαση. Λυπούμε γιατί η... τα σχόλια της Κομισιόν δεν ήταν απόλυτα σαφή. Υπήρχαν πολλές αρνήσεις στη σειρά λέτε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι ωφέλιμη για τους Σαχαραούι. Ε, δηλαδή τι αποδείξεις έχετε ότι όντως είναι ωφέλιμη η συμφωνία αυτή. Συγκεκριμένα να μας πείτε, τι ε, ενδείξεις, αποδείξεις, στοιχεία ζητήσατε υπήρχε στην ε, ημερήσια διάταξη της Δευτέρας και Τρίτης Φεβρουαρίου στην κοινή συνεδρίαση στο Ραμπάτ το θέμα αυτό. Οπότε ρωτώ, τι πληροφορίες λάβατε, τι ερώτημα θέσατε στις μαροκανικές αρχές. Και σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι σας ικανοποίησαν αυτά που λάβατε ως απάντηση. Και επίσης, συμφωνώ με τον κύριο Ρωμέβα, ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τις δύο πλευρέ. πλευρές. Αν δείτε τι λένε οι Σαχαραοί, έχετε, θα δείτε ότι υπάρχει τελείως διαφορετική οπτική. Από την πλευρά τώρα του Κοινοβουλίου, εμείς έχουμε ευθύνη και λόγω αυτής της ε, ασαφούς κατάστασης το Κοινοβούλιο ίσως να πρέπει να δημιουργήσει μια διαρευνητική επιτροπή για να ερευνήσει το θέμα. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό δυνάμει του 226 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε, αν δεν λάβουμε ε, ικανοποιητικές απαντήσεις από την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο μπορεί να δημιουργήσει αυτή την Επιτροπή. Και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το κάνουμε. Και να προσθέσω και κάτι άλλο, ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς την Κομισιόν. Οι εταιρικέ σχέσει και το σχετικό πρωτόκολλο ζητούν από το, από το Μαροκό να δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι ε, συντεταγμένε για τι ληφτικέ ζώνε του Μαρόκου. Μήπω μπορείτε να μα δώσετε αυτέ τι συντεταγμένε των ληφτικών μαροκινών ζωνών. Στη συμφωνία, στο κεφάλαιο 5 ρήτρα 2. Αυτά. Ευχαριστώ. Κυρία Βέστλουντ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω μπορώ να μιλήσω σου ειδικά, έτσι δεν είναι. Είμαι μεταξύ αυτών που, που καταψήφισαν την συμφωνία. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δεν ήμασταν σίγουροι ότι ε, η, συμφωνία ήταν διαρθρωμένη κατά τρόπον ώστε τα ωφέλη να φτάσουν στον πληθυσμό της Δυτικής Σαχάρας. Και δεύτερον, διότι δεν προέβλεπε επουδενή η συμφωνία την δυνατότητα να ακούσουμε τις επιθυμίες των κατοίκων της και των λαών της Δυτικής Σαχάρας. Για αυτούς τους δύο λόγους το κόμμα μου ε, ήταν πεπισμένο ότι η συμφωνία αντίκειται με το διεθνές δίκαιο και πιθανότατα και με τις επιθυμίες των λαών της Δυτικής Σαχάρας. Του λαού της Δυτικής Σαχάρας καλύτερα. Πρέπει να ακούσουμε το λαό της Δυτικής Σαχάρας, αυτό μας το επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Σε ό,τι αφορά την απάντηση της Κομισιόν, με εκπλήσει το γεγονός ότι χρόνια μετά την αρχή της ε, συζήτησης η Κομισιόν λέει ότι δεν έχει αρκετές πληροφορίες. Μα τι κάνετε τόσα χρόνια. Το θέματα αυτά ήταν επίμαχα και συζητούντο για όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ η ίδια έχω πληροφορίες. Υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι του λαού της Δυτικής Σαχάρας που λένε ότι δεν Ακούγεται η φωνή τους σε αυτές τις συμφωνίες. Λοιπόν, γιατί η Κομισιόν ακούει μόνο τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, γιατί δεν ακούτε τον ίδιο το λαό, ο οποίος υφίσταται τα πάνδυνα όλα αυτά τα χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να μην ακούμε τους ανθρώπους και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, όταν σε άλλες περιπτώσεις τις ακούμε σε άλλα μέρη του πλανήτη. Μπορείτε να μου πείτε μια άλλη περίπτωση ε, που μιλάμε μόνο με την κυβέρνηση και όχι με κανέναν άλλον. Είναι δυνατόν αυτό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή τη συμφωνία σίγουρα, αλλά είμαστε πλέον στο 2010. Η συμφωνία ισχύει εδώ και τρία χρόνια και ακόμα δεν έχουμε τίποτα που να μας πείθει ότι θα ωφελήσει το λαό. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Δεν έχει σχέση αυτό με το λαό της Δυτικής Σαχάρας. Έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραβιάζουμε το διεθνές δίκαιο. Δεν είναι αρκετό να λέμε ότι δεν διαθέτουμε αρκετέ πληροφορίες. Πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει και θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε το διεθνές δίκαιο χωρίς να βλέπουμε και να εξετάζουμε τις επιπτώσεις του στα άτομα και στους λαούς. Η Κομισιόν ξέρει τι συμβαίνει και πρέπει να ξέρει τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να μας λέει ότι δεν έχουμε πληροφορίες. Κύριο Στίβενσον. κατανοώ και συμπονώ το λαό της Δυτικής Σαχάρας. Και αν αυτοδιοικούντο, το πρόβλημα θα είχε λυθεί αυτομάτως. Δυστυχώς, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Και ανεξαρτήτως του τι θα θέλαμε, δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις για αυτά τα θέματα. Αυτό συνέβη και με τη Συμφωνία της Γουινέας. όλο και περισσότερο ε, ασχολούμαστε με θέματα που έχουν σχέση με την πολιτική και την εξωτερική πολιτική και, και λιγότερο με την αλία. Κανείς δεν μας λέει ότι αν απο... αχωρήσουμε από την συμφωνία αυτή οι Μαροκινοί δεν θα εκμεταλλευτούν με άλλο τρόπο τα αποθέματά τους χωρίς να ωφελούν πάλι την Δυτική Σαχάρα. Υπάρχουν ε, αντικρώμε απόψει. Άλλοι λένε ότι ωφελείται ο λαό τη Δυτική Σαχάρα, άλλοι, όπω η Κομισιόν, λένε, ε, άλλοι λένε ότι δεν ωφελείται. Η Κομισιόν λέει ότι ωφελείται. Ε, αν όμω εμεί αποχωρήσουμε τη συμφωνία, πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το Μαρόκο δεν θα επιτρέψει στου Ρώσου ή του Κορεάτε να εκμεταλλευτούν αυτά τα αποθέματα. Πώ είμαστε σίγουροι ότι σε αυτή την περίπτωση θα απασχολούνται ε, άτομα, ε, πολίτες της Δυτικής Σαχάρας, πώς θα είμαστε σίγουροι ότι τα αλλιεύματα θα ξεφορτώνονται στη Δυτική Σαχάρα. Δεν θα είμαστε. Πολλές φορές προσπαθούμε να βοηθήσουμε κάποιους και τελικά καταλήγουμε να τους βλάπτουμε. Συνεπώς, το θέμα είναι ένα ε, ζήτημα που απασχολεί τη διεθνή σκηνή, τη διεθνή πολιτική. Εμείς σας παραμείνουμε στη δική μας ειδικεύση, που είναι η αλία. Έχουμε συμφωνία ε, με το Μαρόκο που μας υποχρεώνει ε, να εξασφαλίζουμε πως ε, απασχολούνται άνθρωποι στη Δυτική Σαχάρα, ότι τα λιεύματα ξεφορτώνονται στη Δυτική Σαχάρα κλπ. Και αν μπορούμε να απαιτήσουμε από την Κομισιόν να συλλέξει περισσότερες πληροφορίες για τα ωφελήματα υπέρ του λαού τη Ξαχάρα, αυτό θα ήταν πολύ χρήσιμο. Αλλά δεν νομίζω θα ήταν η σωστή επιλογή να αποχωρήσουμε από την συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Στίβενσον. Έχω ένα μακρύ κατάλογο ομιλητών. Εγώ θα δώσω το λόγο σε όλους βέβαια για να μην με κατηγορήσει, να μην κατηγορήσει κανένα για τίποτα, αλλά δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Κύριο Φερέιρα, παρακαλώ σύντομα για να περάσουμε και στα επόμενα θέματα τη ημερησία διάταξη. Ναι, κυρία Πρόεδρε, θα είμαι σύντομος, γιατί συμφωνώ επί με πολλά από όσα είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι, με εξαίρεση αυτά που είπε ο κ. Στίβενσον. Η απάντηση της ε, Κομισιόν ε, είναι πρώτον ελπίς και δεύτερον αντιβαίνει με τα γεγονότα και τα ε, στοιχεία που έχουμε. Αυτή τη στιγμή το Μαρόκο είναι de facto ε, δύναμη που διοικεί την ε, Σαχάρα κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου. Υπάρχουν ψηφίσματα του ΟΗΕ που καταγγέλουν και καταδικάζουν την εκμετάλλευση των ε, πόρων της Δυτικής Σαχάρας κατά παράβαση των συμφερόντων του λαού και αφαιρώντας τους τα αναπόσπαστα δικαιώματά τους για την εκμετάλλευση των ιδίων πόρων τους. Το γεγονός ότι η Κομισιόν, δεν, ε, το γεγονός ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι ε, ωφελείται ο λαός της Δυτικής Σαχάρας οφείλεται στο ότι μιλάει μόνο με την κυβέρνηση του Μαρόκου. Έχουμε πάρα πολλές αμφιβολίες και γι' αυτό το λόγο είναι αδύνατον να διατηρηθεί συμφωνία με του όρου που ισχύουν αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Στίβενσον, εμεί είμαστε μια πολιτική επιτροπή. Είμαστε πολιτική αλλιώ, αλλά πολιτική επιτροπή. Που τώρα πια έχουμε και διευρυμένε αρμοδιότητε με την νέα συνθήκη τη Λισαβόνα. Συνεπώ, έχουμε ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα μπροστά μα. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε και να πούμε ότι είμαστε τεχνοκράτες δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι αν δεν εκμεταλλευτούμε εμεί τα ε, ελευθερικά αποθέματα τη Δική σαχάρας, θα τα εκμεταλλευτούν κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δεν μπορώ να αγνοήσω ένα τέτοιο μεγέθους πολιτικό πρόβλημα. Δεν πρόκειται να το κάνω εγώ. Και τελειώνω με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω, λάμβαντας υπόψη την κατάσταση, ότι είναι επίγον να διευκρινιστεί η θέση της Κομισιόν και να πρέπει να ζητήσουμε πιο ασφαλή και πιο καθαρά στοιχεία από την Κομισιόν. Θέλουμε να γίνει μία επίσκεψη στο Μαρόκο με επισκέψεις στους λιμένες της Δυτικής Σαχάρας. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας μπορεί να την οργανώσει αυτή την επίσκεψη. Θα μας επιτρέψει να γνωρίσουμε καλύτερα από κοντά την κατάσταση και τότε θα σταθμίσουμε Ε, την ε, συμμετοχή μας με τους τρόπους με τους οποίους μας προτείνετε. Ευχαριστώ. Κυρία Άντρες Βαρέα. Βρισκόμαστε στην Επιτροπή Αλίας και συζητούμε μια συμφωνία Αλίας, αλευτική συμφωνία. Ε, η κυριαρχία την κυριαρχία δεν την έχει το Μαρόκο επί της ε, Δυτικής Σαχάρας. Έτσι. Ε, αλλά έχει τη δικαιοδοσία. Δικαιοδοσία σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα διαχείρισης το Μαρόκο επί της Δυτικής Σαχάρας. Η συμφωνία στις 2 Φεβρουαρίου αναθεωρήθηκε, το είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, με πρόβλεψη προ, πρόσθετων δραστηριοτήτων υποστήριξη του τομέα. Ίσως δεν ήταν αρκετό, θα προβλεφθούν και άλλα πράγματα, αλλά σίγουρα ίσως αγνοούμε, όπως και σε άλλες συμφωνίες, το κατά πόσον έχει εφαρμοστεί και με ποιο τρόπο. Όμως, ζητήθηκε μια τροποποίηση, <clears throat> έγινε μια τροποποίηση Αν θέλουμε, μπορούμε να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά προκειμένου να ζητήσουμε την αναστολή, χρειάζεται να έχουμε πολύ περισσότερα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουμε εμείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή τέτοιου είδους αποχώρηση, αν υπάρχουν προβλήματα, αυτό θα πρέπει να γίνει φανερό από συγκεκριμένα στοιχεία. Μιλούμε για την αλία, μιλούμε για την δικαιοδοσία και όχι για την κυριαρχία του Μαρόκου. Κυρία Μπιλμπάου. Η συμφωνία είναι υπογεγραμμένη, έχει συναυθεί. Εγώ πριν φτάσω στο Κοινοβούλιο υποστήριζα πάντοτε την, το δικαίωμα ε, αυτοδιαχείρισης της ε, Δυτικής και τα συμφέροντα του λαού τη Δυτικής Σαχάρας ε, αλλά θα ήθελα να ζητήσω διαφάνεια από την Επιτροπή και απαιτώ ως μέλος αυτής της Επιτροπής Αλίας από την Κομισιόν μια έκθεση με την αξιολόγηση του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων αυτής της συμφωνίας. Και ζητώντας διαφάνεια, ζητώ μια λεπτομερή έκθεση για τα ωφέλη τα οποία άντλησε ο λαός της Δυτικής Σαχάρας από την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Το ίδιο και ο λαός του Μαρόκου. Η νομική υπηρεσία μας είπε ότι πριν τον Αύγουστο πρέπει να καθορίσουμε τη θέση μας, γιατί η συμφωνία λύγει το 2011. Έχω την εντύπωση ότι ε, μιλάμε όλοι με υποθέσεις γιατί λείπουν οι πραγματικές πληροφορίες. Συνεπώς, ήρθε η στιγμή να ζητήσουμε την απαραίτητη διαφάνεια, να απαιτήσουμε την απαραίτητη διαφάνεια από την Κομισιόν. Γιατί με τη συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξαν και οι δικές μας αρμοδιότητες. Από εδώ και πέρα θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε αναξαρτήτως της θέσης μας για, την, για το πρόβλημα της Δυτικής Σαχάρας θα έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογούμε την κατάσταση και να λαμβάνουμε θέση. Για να λάβουμε όμως αυτή τη θέση η Κομισιόν θα πρέπει να μας υποβάλει μια διαφανή, πλήρη ε, και λεπτομερή έκθεση έτσι ώστε μέχρι τον Αύγουστο να έχουμε χρόνο να καθορίσουμε τη θέση μας αναλύοντας την κατάσταση αντικειμενικά προκειμένου να, λάβει άποψη, να έχει άποψη για το, το μέλλον της συμφωνίας. Ευχαριστώ. Κύριος Μιλάνα. Η παρέμβαση της κυρίας Μπιλμπάου με βρίσκει σύμφωνο. Και εγώ τα ίδια ήθελα να πω αντιμετωπίζουμε μια συμφωνία που ουσιαστικά είναι εμπορική συμφωνία. Όσον αφορά το, το νόμο, αν η προσέγγιση που ακολουθούμε ως Ευρώπη έναντι αυτών των συμφωνιών είναι απλώς εμπορική, έχει δίκιο ο κύριος Στίβενσον. Αλλά κατά την άποψή μου δεν είναι εμπορική συμφωνία. Τουλάχιστον αλληλευτικές συμφωνίες δεν μπορούν να είναι αποκλειστικά εμπορικές συμφωνίες. Ή δεν μπορεί να είναι μόνο να ερμηνευτεί εμπορικά από πλευρά αγορά Συμφωνώ με αυτό που είπε η συνάδελφο. Αν ακολουθήσουμε αυτή την προσέγγιση, δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να συζητήσουμε πλέον. Διότι η αγορά ρυθμίζει αυτέ τι σχέσει. Κάνουμε τι αλευτικές συμφωνίε μα βολεύει. Εγώ επέστρεψα από ταξί στη Μαυριτανία. Πήγα με την αντιπροσωπεία για το Μαγκρέμπ και έχουμε μεγάλη αλληλευτική συμφωνία με τη Μαυριτανία. Και έχει δικτατορία η Μαυριτανία. Όταν ζητήσαμε από τους υπουργούς και τους άλλους να μας πούν ποια είναι τα ωφέλη για τους τοπικούς πληθυσμούς, μας είπαν κανένα όφελος. Τα χρήματα πάνε στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση τα χρησιμοποιεί. Δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών της Μαυριτανίας και του Πρωθυπουργού. Πιστεύω λοιπόν ότι από αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να αντιλήσουμε κάποια αξιολόγηση. Και αυτή η αξιολόγηση ποια είναι. Επιλέγουμε και θέτουμε τι ελευθερικέ συμφωνίε σαν κάτι εμπορικό, σε εμπορικό πλαίσιο, τότε τελείωσε ο αγώνα. Αλλά αν θέλουμε να παίξουμε κοινοβουλευτικό ρόλο, δεν μπορεί να έρχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προσβάλλομαι από τι δηλώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γνωρίζω δεν υπάρχει, δεν μπορώ να συμπεράνω ότι μεταφέρονται ωφέλη προς τους ντόπιου πληθυσμού της Σαχάρας. Αυτό δεν είναι απάντηση και συμφωνώ με την κυρία Μπιλμπάου που λέει πρέπει κατεπηγόντως Έχουμε μέχρι το 2011, έχουμε χρόνο. Κατεπηγόντω, μια έκθεση Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπομειστεί την ευθύνη και να μα πει άπαξ διαπαντό αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν οι κάτοικοι τη Σαχάρα, Σαχράουι, Δηλαδή ούτε Σαχράουι, ούτε ο λαός της Σαχάρας, ούτε οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Σαχάρας υπάρχουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κάνει αυτή τη δήλωση, μπορούμε να κάνουμε συμφωνία χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορεί να συνεχίσει να λέει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει το θέμα για τη δυτική Σαχάρας, ότι θα ρυθμιστεί στον ΟΗΕ και σκασίλα μας εμάς. Θα πρέπει να έρθει η κυρία Άστον εδώ και στην Επιτροπή Αλίας. Διότι η Επιτροπή Αλίας δεν είναι μια επιτροπή που έχει βουλευτές που είναι μόνο είναι έξυπνα άτομα τα μέλη της ε, Επιτροπής Αλίας έχουν ευφυΐα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί προ όφελο τη της κοινότητάς μας. Κυρία Βαντούστ. Ε, Κυρία Ράντουστ. Θα συμφωνήσω. Και εγώ θεωρώ ότι είμαστε πολιτική επιτροπή. Εγώ είμαι πολιτικός και δεν είμαι εδώ σε εκπρόσωπος κάποιου εμπορικού οργανισμού πρέπει να λάβω πολιτικές αποφάσεις και θα τις λάβω δυνάμει της ε, κοινωνικής δικαιοσύνης και της βιωσιμότητας. Όταν συνάπτουμε μια συμφωνία αλληλευτική, θεωρώ ότι όλοι οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από αυτή. Και το... Ε, οι καιροί πέρασαν που εμείς εδώ ήμασταν μόνο οι καλοί, οι Ευρωπαίοι, Ήδη είδαμε τι έχει γίνει και με τη συμφωνία της ε, Γουινέας. Αυτά έτσι ως αρχικές παρατηρήσεις. Πρέπει να πω ότι αισθάνομαι λίγο προσβεβλημένη, όπως ο συνάδελφος Μιλάνα. Νομίζω ότι ε, είμαστε λίγο υπερόπτες. Ξέρουμε ποιο είναι, το θέμα στην ημερήσια διάταξη και λέμε με τρεις φράσεις «Α, εγώ δεν ξέρω περισσότερα, ξέρω μόνο αυτό» ε, νομίζω ότι η Κομισιόν θα έπρεπε να μας δώσει κάτι παραπάνω. Αν είναι τώρα κάποιο σημείο το οποίο ε, ετέθη πολύ πρόσφατα στην ημερήσια ε, διάταξη, περιμένω να ερευνηθεί το θέμα περαιτέρω και να λάβουμε πληροφορίες. Δεν έχουμε λάβει τίποτα, οπότε ζητώ πληροφορίες άμεσα γιατί εγώ εξελέγην για να διακόψω αυτή την συμφωνία. Αν δεν λάβω καλύτερες ε, πληροφορίες, θα φροντίσω στις, ε, να μην ε, ανανεωθεί η συμφωνία αυτή στις 26 Αυγούστου. Μιλούμε για ανθρώπους που δεν ακούγεται η φωνή τους και οι άνθρωποι στο Μαρόκο επίσης ζουν σε μια περίεργη κατάσταση. Τώρα για, την, ε, ε, για το να δημιουργήσουμε αυτή την ε, διαρευνητική επιτροπή ίσως να πρέπει να το συζητήσουμε με την ομάδα μου για να δούμε κατά πόσο μπορεί αυτό να γίνει άμεσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά και εγώ είμαι συγκλονισμένος με την απάντηση της Επιτροπής. Ε, μη ύπαρξη πληροφοριών δεν μπορεί να είναι μια απάντηση σε αυτήν την Επιτροπή. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η κυρία Ροντάς. Ε, ταυτίζομαι απόλυτα με την θέση, όπως και με τη θέση των συναδέλφων, όπως εκφράστηκε μέχρι στιγμής. Πραγματικά ε, νιώθω συγκλονισμένος από αυτά που ακούσαμε σήμερα και αναρωτιέμαι αν η Επιτροπή ε, έχει κάποιες, κάποιες αποδείξεις τουλάχιστον για, τις, για το ότι φτάνουν κάποιες από τις ωφέλεις της συμφωνίας του Σαχαράουι και αν η Επιτροπή έχει αναζητήσει αυτές τις αποδείξεις. Ε, κατά τα άλλα παραμένω ακριβώς στην, ε, στη γραμμή ακριβώς όπως τα, έθεσε η κυρία Ροντάστ. Πραγματικά, αν δεν έχουμε άμεσα αυτές, τις βασικές αυτές πληροφορίες και αν δεν έχουμε μια, άμεσα μια ε, πιο συνεπή απάντηση από την Επιτροπή, ε, και εγώ θα ταχθώ υπέρ της διακοπής αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ κύριε Αρσένη. Να πω και εγώ τη γνώμη μου. Καταρχήν να σας πω ότι η σημερινή συνεδρίαση είναι ανοιχτή. Δεν είναι και κλεισμένο το θυρών. Θα κάνω μια πρόταση στο τέλος ε, να οργανώσουμε μια συνεδρίαση από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κλεισμένων των θυρών. Είναι προφανές ότι ε, με παρουσία ε, κοινού ορισμένα θεσμικά όργανα δεν μπορούν να μιλήσουν με την ελευθερία που θα είχαν αλλιώς. Σας το λέω αυτό για να καταλάβετε ποιο είναι το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Ίσως καλύτερα θα ήταν να οργανώσουμε μια συνεδρία κλεισμένων των θυρών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερον, Εγώ συμφωνώ με τον κύριο Στίβενσον, παρόλο που πολλοί από εσά διαφωνείτε. Ε, το θέμα της Δυτικής Σαχάρα είναι πολιτικός ε, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχουμε μπροστά μας. Ε, δηλαδή πολύ πιο πλατή από την ε, Συμφωνία. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για να το χειριστούμε. Τώρα, για τα νομικά ζητήματα που μας ανέφερε ο κ. Πάσος. Θα ήθελα να υποβάλω τι εξή ερωτήσει προ τον κύριο Πάσο και μετά μία ερώτηση προ την Κομισιόν. Όταν μιλούμε για του τοπικού πληθυσμού, ε, άλλο καταλαβαίνει η Ευρώπη γι' αυτό, άλλο καταλαβαίνουν οι Μαροκινοί. Πρέπει να δούμε ποια είναι, ποιος είναι ο τοπικός ε, πληθυσμός για να δούμε αν ωφελείται. Γιατί το Μαρόκο θεωρεί τοπικό πληθυσμό κάτι διαφορετικό από αυτό που θεωρούμε εμείς. Συνεπώς, θα πρέπει να είμαστε σαφείς στη νομική ορολογία που χρησιμοποιούμε. Δεύτερον, όταν μιλάτε για επαρκή ωφέλη, τι σημαίνει ακριβώς επαρκή ωφέλη. Όλα τα ποσά που πληρώνονται για την αλληλευτική συμφωνία θα έπρεπε να φτάνουν στο λαό ή ένα κομμάτι όλη η ενα κομματι όλοι η αναπτυξιακή βοήθεια που δίδεται. Δεν καταλαβαίνω πώς αποφασίζουμε αν ε, είναι επαρκέ επαρκές το όφελος. Γιατί η συμφωνία έχει δύο τμήματα. Το εμπορικό τμήμα και το τμήμα αναπτυξιακής βοήθειας. Συνεπώς πρέπει να ξέρουμε την απάντηση για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις πληροφορίες της Κομισιόν ή του Μαρόκου. Τρίτη ερώτηση που μάλλον θα μου την απαντήσει καλύτερα η Κομισιόν. Πρέπει να τη θέσω όμως. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αλευτική Συμφωνία έχει ένα εμπορικό τμήμα, όπως είπα, και ένα τμήμα αναπτυξιακό. Με κειμενόμενα ποσοστά, όλες οι αλευτικές συμφωνίες έχουν δύο κομμάτια. Σε άλλες συμφωνίες είναι 80% το ένα και 20% το άλλο, σε άλλες 70-30% κλπ. Όλες οι αλευτικές συμφωνίες έχουν την ίδια μορφή. Αυτό που ισχύει όμως είναι ότι το κομμάτι για την αναπτυξιακή συνεργασία ε, εστιάζεται αποκλειστικά στην αλία. Δηλαδή, τα ποσά τα οποία δίδονται στο πλαίσιο αυτού του κομματιού, αυτού του κλάδου, πρέπει να φτάσουν στην αλία. Όχι να χτίζονται νοσοκομεία, για παράδειγμα. Συνεπώ, το όφελο που θα πρέπει να αντλεί ο τοπικό εισαγωγικά πληθυσμό τη Δυτική Σαχάρα θα πρέπει να είναι όφελος υπέρ του αλλιευτικού τομέα. Όχι νοσοκομεία ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή, έτσι. Τα χρήματα που φτάνουν μέσω της αλλιευτικής συμφωνίας πρέπει να ωφελούν τον αλλιευτικό τομέα. Συνεπώς, ας υποθέσουμε ότι τοπικός πληθυσμός είναι ο πληθυσμός ο οποίος εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης δεν μπορεί να επωφεληθεί του δεύτερου αυτού κομματιού. Τι θα συμβεί τότε. Τέταρτον, εγώ ήρθα από το Μαρόκο πολύ πρόσφατα. Ξέρω ότι στο λιμάνι της Δάκλα, στη Δυτική Σαχάρα, το Μαρόκο προβλέπει ε, διάφορες υποδομές και την ανάπτυξη του λιμανιού του Ελαϊγιούν. Συνεπώς ένα κομμάτι της ε, αναπτυξιακής βοήθειας που δίνουμε εμείς στο Μαρόκο φτάνει στη Δυτική Σαχάρα. Συνεπώς τι θεωρούμε ότι είναι επαρκές όφελος. Και μετά σας είπα πρέπει να δούμε το κατά πόσον αυτή η αναπτυξιακή βοήθεια ε, φτάνει τον αλληλευτικό τομέα και κατά πόσο είναι λογικό ορισμένοι οι οποίοι δεν ασκούν αλληλευτική δραστηριότητα στη Δυτική Σαχάρα να μην βλέπουν όφελος από αυτή τη συμφωνία. Μετά να σχολιάσω και κάτι που ο κ. Μιλάνα. Σε όλες τις συμφωνίες το εμπορικό κομμάτι η οικονομική αντιστάθμιση που αφορά το εμπορικό κομμάτι ε, δεν απαιτεί αιτιολόγηση από την δικαιούχο χώρα. Αυτό που χρειάζεται να αιτιολογηθεί είναι η χρήση των πόρων για, την αναπτυξιακή, ε, για το αναπτυξιακό σκέλος. Και γι' αυτό λόγο υπάρχουν και οι μικτές επιτροπές στη συγκεκριμένη περίπτωση το, με το Μαρόκο, όπου ε, η αντίστοιχη χώρα δικαιολογεί τις δαπάνες κλπ. Θα δώσω το λόγο σε δύο ακόμα ομιλητές και μετά αν θέλετε μπορούμε να προτείνουμε μια ε, συνάντηση και κλεισμένων των θυρών με την ε, Κομισιόν. Κύριος Πάσος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν με εκπλήσει, δεν με εκπλήσουν τα ερωτήματα που θέσατε. Είναι πολύ σημαντικά. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μερικές ε, απαντήσεις. Δεν έχω όμως όλες τις απαντήσεις που ζητάτε. Δεν έχω αρκετά στοιχεία. πρώτη σα ερώτηση ήταν πολύ σημαντική. Πώ ορίζεται ο τοπικό πληθυσμό, Είπατε ότι υπάρχουν δύο πλευρές που βλέπουν διαφορετικά αυτή την έκφραση. Αυτό που μπορώ να σα πω εγώ πριν απαντήσω στην ερώτηση είναι ότι μπορώ να σα παραπέμψω στην κατάσταση που ανεξαρτήτως των πολιτικών του Μαρόκου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, των σχέσεων, αλευτικών σχέσεων με το Μαρόκο κλπ. Το γεγονός είναι ότι η Δυτική Σαχάρα ε, δεν είναι αυτοδιοικούμενη περιοχή σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Και αυτό δεν αμφισβητείται. Επίσης, ε, εκκρεμεί επίλυση του προβλήματος της Δυτικής Σαχάρας αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό το μήνα έγινε μια συνάντηση στη Νέα Υόρκη για τη Δυτική Σαχάρα. Και σας παραπέμπω σε ένα δελτίο τύπου της 12 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα προέρχεται από την Υπηρεσία Ειδήσεων του ΟΗΕ που αναφέρεται σε αυτές τις συνεχιζόμενες συζητήσεις. Δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι ένα πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται. Το δελτίο τύπου λέει ότι τα μέρη ε, ε, συμμετείχαν σε μια διήμερη συνάντηση στη Νέα Υόρκη και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους, την προσήλωσή τους να συνεχίσουν διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Οι προτάσει των δύο μερών ξαναπαρουσιάστηκαν και ξανασυζητήθηκαν. Στο τέλος της συνεδρίασης, καμία από τα δύο μέρη δεν είχε δεχτεί τις προτάσεις του άλλου. είπε ο κ. Ρο, προσωπικό απεσταλμένο του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση έγινε με σοβαρότητα, ε, φιλικότητα και αμοιβαίο σεβασμό. Συνεπώ, δεν θα βρει λύση η δική σα Επιτροπή. Το θέμα εκκρεμεί στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτοί θα βρουν τη λύση. Αλλά ο ντόπιο πληθυσμό δεν ορίζεται. Αν υπάρχουν δύο ερμηνείε, θα πρέπει να τι λάβουμε και τι δύο υπόψη. Εγώ δεν μπορώ να σα πω ποιο είναι ο ντόπιο πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά τα ωφέλη. Σίγουρα υπάρχει ένα κομμάτι που είναι εμπορικό και ένα κομμάτι που είναι ε, ε, αναπτυξιακό. Σίγουρα ε, το εμπορικό θα πρέπει να φτάνει στον αλληλευτικό τομέα. Είναι μια κλαδική συμφωνία, αλλά είναι όμως και συμφωνία αναπτυξιακή. Συνεπώς λέτε, αυτά τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, για νοσοκομεία ή για δρόμους κλπ. Θα πρέπει να φτάσουν στον αλληλευτικό τομέα. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Είναι σίγουρο ότι η συμφωνία είναι αλληλευτική συμφωνία και καταρχήν ε, τα κονδύλια που δίδονται αφορούν την αλευτική πολιτική. Όμως το γεγονός είναι πως το Μαρόκο είναι το έτρο συμβαλόμενο μέρος και η συμφωνία αυτή αφορά μια περιοχή η οποία ε, δεν εμπίπτει στην επικράτεια του Μαρόκου σύμφωνα με το Εθνές Δίκαιο. Λοιπόν, ε, ε Όποιο και αν είναι ο ντόπιο πληθυσμό θα πρέπει να ωφελείται. Αν θα είναι μόνο ο αλευτικό τομέα ή όχι, ε, γι' αυτό δεν είμαι σίγουρο. Δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι το Μαρόκο μπορεί να πει το εμπορικό κομμάτι δεν έχει σχέση με εσά, Δυτική Σαχάρα. Οι δέσμευση που έχουν σύμφωνα με το διεθνέ δίκαιο είναι ότι θα πρέπει να ωφελείται ο τοπικό πληθυσμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον. Κάποια μέλη μίλησαν και για ενδεχόμενη αναστολή της συμφωνίας. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση και πάλι έχουμε ελπίς πληροφορίες σε κάθε περίπτωση αν υπάρξει πρόβλημα η κοινή επιτροπή θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες της η μεικτή επιτροπή θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες της γιατί σύμφωνα με την συμφωνία στο άρθρο 10 αναφέρεται πως η μεικτή επιτροπή αν υπάρχει πρόβλημα είναι ο, η Επιτροπή που έχει την ευθύνη του φιλικού διακανονισμού οποιονδήποτε διαφορών προκύψουν. Δεν ξέρω αν κάνουν κάτι τέτοιο. Α, δεν έχω πληροφορίε. Ζητώ συγγνώμη δεν μπορώ να απαντήσω όλες τις ερωτήσεις ε, ε, με τρόπο απολύτως ακριβή όπως θα θέλατε, αλλά δεν έχω και εγώ όλες τις πληροφορίες που θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Ο κ. Φοντάνα τελευταίος, έτσι κι αλλιώς θα γίνει συνάντηση και κλεισμένο των θυρών. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Για να ολοκληρώσω αυτά που προανέφερα, είπα ότι δεν είχαν πληροφορίες που να δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ωφέλη. Έχουν πληροφορίες για ωφέλη για τη Δυτική Σαχάρα. Σαν συνέπεια των αλληλευτικών δραστηριοτήτων, πράγματος χάρη, υπάρχουν εκφορτώσεις αλλιευμάτων στα λιμάνια του Νότου αυτό δημιουργεί οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση. Ξέρουμε ότι προσλαμβάνονται ναυτικοί επιτόπου και ιδιωτικές επενδύσεις δόθηκαν στην τάχλα και δημιουργούν οικονομικές δραστηριότητε. Αυτά είναι συνέπειες των οικονομικών δραστηριοτήτων. Τώρα, όσον αφορά την υποστήριξη του τομέα, Δηλαδή το κομμάτι της συμφωνίας που είναι πρόγραμμα με συγκεκριμένε δραστηριότητε που εντάσσονται στη Γενική Συμφωνία δραστηριότητε, θα ξέρετε την τελευταία τριετία υπάρχουν κατηγορίες τομεακών ενισχύσεων προχώρησαν περισσότερο και άλλοι τομεί δεν έχουν καλυφθεί τόσο πολύ. κατηγορίε που στηρίχθηκαν περισσότερο είναι η κατάρτιση. Και εντό τη κατάρτιση Ξέρουμε από τις συζητήσεις που έγιναν στην Μικτή Επιτροπή ότι υπήρξε υποστήριξη για το κέντρο της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων στον τομέα της αλίας στην Τάχλα και το Τεχνικό Ινστιτούτο για Αλληλία στον Ταγιούγκ. Και πιστεύουμε ότι αυτού του είδους οι δραστηριότητες στην Τάχλα και στην Αγιούγκ ε, αυτές οι δραστηριότητε ωφελούν τους ντόπιου πληθυσμούς του των λεχθέντων στη Μικτή Επιτροπή όπως σας προανέφερα Ζητήσαμε και άλλες πληροφορίες όσον αφορά τα ωφέλη που απορρέουν τη συμφωνία και αυτό φαίνεται και από τα συμπεφωνημένα πρακτικά της Επιτροπής και προσβλέπουμε στις πρόσθετες πληροφορίες και όταν τις λάβουμε θα τις μοιραστούμε με την Επιτροπή σας όπως πρότεινε και η κυρία Φράγα. Ευχαριστούμε τον κύριο Φοντάν, ευχαριστούμε τον κύριο Πάσος θα διοργανώσουμε μια συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών έτσι ώστε η Κομισιόν να μας ενημερώσει πιο λεπτομερώς για τη συμφωνία σύμπραξη με το Μαρόκο. Κλείνουμε το σημείο 6 μέσης διάταξης, περνάμε στο σημείο 7. Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλλιευμάτων για τον, τον Τούνους Τίνους. Ε, εισηγητής ο κ. Ε, Ρωμέβα Ιρουέδα. Κύριε Ρωμέβα. Το θέμα αυτό φαίνεται τεχνικό και είναι, αλλά έχει και μια σημαντική πολιτική διάσταση. Ιδιαίτερω εξαιτία τη ε, απόφαση που πήρε το Κοινοβούλιο πριν μερικέ μέρε και χτε ε, η απόφαση, εξαιτία τη Κομισιόν που σύστησε να υποστηρίξουμε την πρόταση του Μονακό στην Τόχα προκειμένου να περιληφθεί ο ερυθρό τόνο στο πρώτο παράρτημα των απειλούμενων ειδών. Υπάρχουν δύο διαστάσεις αυτήν την έκθεση λοιπόν. Μία είναι η τεχνική που έχει σχέση με την τροποποίηση του ισχύοντος συστήματο, κοινοποίηση των αλλιευμάτων. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσαρμοστεί στις αποφάσεις που ελήφθησαν στην συνέδριαση του Ρεσίφε της ΙΚΑΤ τον, το περασμένο φθινόπωρο και αυτό έχουμε κάνει με την έκθεση. Κάνουμε δηλαδή μια τεχνική μεταγραφή των συστάσεων που θα μας ε, επιτρέψει να βελτιώσουμε έτσι περαιτέρω την ε, πληροφόρηση για τα αλλιεύματα και για τις μεταφορές τις μεταβιβάσεις καλύτερα ε, αυτών των αλλιευμάτων ε, και να προσαρμόσουμε την κατάσταση στα ισχύοντα στην ΙΚΑΤ. Υπάρχει μια σειρά τροπολογιών μέσω των οποίων ε, επιφέρουμε αυτές τις ε, αλλαγές, τις προσαρμογές. Σας καλώ επίσης να διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση για να καταλάβετε καλύτερα το ιστορικό του θέματος. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την τεράστια σημασία την τεράστια αξία αυτού του εγγράφου, όχι μόνο για τα αλλιεύματα ερθρού αλλά και για την βελτίωση της διαφάνειας και του ελέγχου ε, σε ό,τι ε, αφορά την ε, παράνομη αλία. Γι' αυτό το λόγο θα συζητηθεί το ζήτημα αυτό ε, και για τη... Α, οι, δύο τροπολογίες όμως ε, είναι ε, πιο πολιτικές και προκύπτουν εξαιτίας την συζήτηση για τον τελευταίο ημερών και των αποφάσεων των τελευταίων ημερών για την συμπέληψη του Ερθού τόνου στην ΣΥΤΕΣ. Έχουν ως σκοπό να πούν ότι η αναθεώρηση αυτού του εγγράφου θα προσαρμογιστεί ε, στην έκβαση ε, των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα το Μάρτιο. και αν είναι, όποια και αν είναι αυτή η έκβαση. Όποια και αν είναι αυτή η έκβαση θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Συνεπώ, προτείνω να διατηρήσουμε αυτή την διατύπωση ανάλογα με το ποια θα είναι η κατάληξη των συζητήσεων στις ΣΥΤΕΣ με αυτόν τον τρόπο το έγγραφό μας θα είναι πάντα επίκαιρο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ε, απ' την άλλη μεριά, μια και είναι η Κομισιόν εδώ, θα ήθελα να υποβάλω μια σειρά ερωτήσεων σχετικά με την, το τεχνικό σκέλος της, ε, του εγγράφου. Τι εξής ερωτήσεις. Πρώτον, η ερώτησή μου αφορά και το Συμβούλιο. Δεν ξέρω αν είναι παρόν το Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει είναι ανοιχτή η ερώτηση. Αν δεν πάρουμε απαντήσει σήμερα μπορούμε να ζητήσουμε και γραπτές απαντήσεις. Στο πλαίσιο της συνεδρίας ομάδας εργασίας για την ε, Αλία, περασμένη εβδομάδα, ε, προέκυψαν μια σειρά ανησυχιών ή απορριών από τη γαλλική και ιταλική κυρίω ε, αντιπροσωπεία σε ό,τι αφορά τις ε, απαιτήσει των ιαπωνικών αρχών σε ό,τι αφορά θέματα εισαγωγής. Ειλικρινά λέω ότι δεν ξέρω σε τι ακριβώς βασίζονται αυτές οι ανησυχίες. Θα ήθελα να διευκρινιστεί και θα ήθελα να ρωτήσω σε τι βασίζεται η Ιαπωνία κάθε φορά για την, ε, την επιβολή μέτρων περιορισμού των εισαγωγών ερθρού τόνου. Δεύτερον, δεύτερη ερώτηση προς την Κομισιόν. Έχει σχέση με τις ζώνες της αλίευσης. Η ζώνη αλίευσης του ερθρού τόνου είναι πολύ μεγάλη γιατί περιέχει και το, Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο. Συνεπώς, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να καθορίσουμε αλλιευτικές ζώνες πολύ πιο περιορισμένες. Γιατί? Για να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στα στοιχεία αυτών των αλλιευμάτων. πρέπει να λάβουμε υπόψη το ρόλο των ε, ηλεκτρονικών ε, logbooks ε, μητρώων που τηρούνται για τον έλεγχο. Τελευταία ερώτηση προς την Κομισιόν πάλι. Σε σχέση με τη χτεσινή απόφαση. Ενημερωθήκαμε μέσω των ΜΜΕ και στην συνέντευξη τύπου, αλλά δεν έχουμε γραπτό στην απόφαση της Κομισιόν. Υπάρχει αυτό το έγγραφο. Έχει καταγραφεί η απόφαση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την πρόταση της ε, Επιτροπής να συμμεριθεί ο έρθρος τόνος στην ΣΥΤΕΣ. Θα θέλαμε, αν υπάρχει ένα τέτοιο έγγραφο, να μας το προωθήσετε. Ευχαριστώ. Η τηλεόραση των Κανάριων νησιών ε, θέλει να μπει και να κινηματογραφήσει. Αν δεν διαφωνείτε, το επιτρέπουμε. Ωραία. Δίνω το λόγο στον εαυτό μου, μια και δεν το ζητάει κανένα άλλο. Διάβασα, κύριε Ρωμέβα, ε, πολύ καλά την έκθεσή σα και την αιτιολογική έκθεση. Θα ήθελα να κάνω τι εξή παρατηρήσει. Καταρχήν, δύο τροπολογίε, 7 και 44, σχετικέ με τι ΣΥΤΕ. Ε, η θέση σα διαφέρει από αυτήν άλλων μελών μεταξύ των οποίων και τη δική μου. πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ε, ακολουθήσουμε τις επιταγές της ΣΥΤΕΣ, όχι, αντιθέτως. Για τις άλλες τροπολογίες, ε, μπορεί βέβαια να μην, διάβασα, διάβασα καλά, αλλά έχω την εντύπωση πως ερμηνεύεται πιο περιοριστικά την σύσταση της ε, ΙΚΑΤ που έγινε δεκτή στο Ρεσίφε. Δηλαδή δεν διαφωνώ με την ουσία, αλλά νομίζω ότι ερμηνεύεται αυτή τη σύσταση πιο περιοριστικά μερικές φορές. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε γιατί δεν το μπορώ να το συμπεράνω να το καταλάβω από την αιτιολογική έκθεση. Ίσως ε, προσωπικά θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε μερικές τροπολογίες. Έχουμε τη 16, 17 και 18 με τις οποίες συμφωνώ ε, γιατί μεταγράφεται κατά λέξη αυτό που εγκρίθηκε. Παρόλο ότι στις 18 αντί για τις 15 μέρες που αναφέρει στις σύσταση, έχετε βάλει 8. Μπορεί να βάλει περισσότερο 8 αλλά δεν ξέρω γιατί βάλετε 8 αντί για 15. <clears throat> Θα ήθελα να μου το εξηγήσετε πάντως. Υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τη σύσταση, ορισμένες μικρές και ορισμένες πιο μεγάλες. Ε, δεν καταλαβαίνω αυτές τις αποκλήσεις. Βλέπω ότι οι συνάδελφοι γενικώ δεν ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτή την γνωμοδότηση, αλλά γι' αυτό λόγο ενδεχομένω διμερό θα μπορούσατε να μου εξηγήσετε αυτέ τι αποκλήσει. Τώρα για την αιτιολογική έκθεση. Δεν συμφωνώ με τις τελικές παρατηρήσεις, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Κάνετε μια ερμηνεία ενός τμήματος των όσων ελέγχθησαν στην Επιστημονική Επιτροπή της ΕΚΑΤ ε, και στον ΦΑΟ. Ε, δεν καταγράφεται και τις άλλες απόψεις, γιατί, για παράδειγμα, ε, για το θέμα του 15%, του περίφημου 15%, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το προσωπικό μου σχόλιο. Αυτά ε, ε, θα ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο καλύτερα ε, για να καταλάβω σε βάθος την σα. Και σα λέω, εγώ το, τη διάβασα πολύ, προσεκτική, πολύ προσεκτικά, από το α μέχρι το ω, ε. το έχω δουλέψει, έχω, κάνει το, έχω μάθει το μαθημά μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που ετέθησαν Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τι ανησυχίε που εξέφρασαν κάποια κράτη-μέλη λόγω των απαιτήσεων τη Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία ως σημαντική δύναμη εισαγωγική είναι γνωστή διότι επιβάλλει στα άλλα μέρη στον τομέα της αλληλείας, του εμπορίου, απαιτήσει απαιτήσει που αφορούν τα προσεισαγωγήν εμπορεύματα στην αγορά της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία προσπαθεί να προβλέψει, να προδικάσει το ρυθμιστικό, ε, τον χαρακτήρα των προϊόντων που θα μπουν στην αγορά, ώστε να επιτρέψει στους εμπερευόμενους της να αγοράσουν και να επαναπολύσουν με την ησυχία τους τα προϊόντα. Αυτή είναι μια σταθερή θέση που μπορεί να δημιουργεί κάποιες ανισορροπίες μεταξύ του επιμερισμού των ευθυνών στις χώρες σημαίας, στις χώρες μεταποίησης ενδεχομένως και στις χώρες της αγοράς. Η αγορά είναι που τελικά ρυθμίζει τις αληφτικές δραστηριότητε. Αυτό πρέπει να γίνεται, αυτό ουσιώδες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις πρωτοβουλίες της όσον αφορά την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας υποχρεούται να φροντίσει ούτως ώστε οι ευθύνες να μοιράζονται. Αναλογικά να μοιράζονται σε όλους τους εμπλεκόμενους. Σε αυτή την πρόταση. Λοιπόν, σε αυτή την πρόταση είναι πολύ σημαντικό αν οι χώρες σημαίας φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των σκαφών τους να ελέγχουν κατά πόσο είναι νόμιμες οι δραστηριότητες και να μην επικυρώνουν τα έγγραφα αλληλείας εάν δεν είναι σωστές οι δραστηριότητες. Εξίσου σημαντικό είναι και οι χώρες εισαγωγής να μπορούν να υπομισθούν τις ευθύνες τους στα πλαίσια της όλης ρύθμισης. Και γι' αυτό τα κράτη-μέλη εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Λοιπόν, και αυτός ο μηχανισμός για τα αλλιεύματα λαμβάνει υπόψη τη συνεργασία με τα κράτη αγωγής για να πετύχουμε τους στόχους τους επιθυμητούς. Τώρα, όσον αφορά τον ακριβέστερο ορισμό των διαφόρων ζωνών αλλίες εκεί που ε, αλλιεύεται ο ρηθρός τόνος. Υπάρχουν δύο μεγάλες ζώνες. Το να κάνουμε πιο ακριβή διαίρεση των ζωνών αυτό θα ήταν, θα αρμοδιότητα άλλου φορέα, περιφερειακού, που καθορίζει τις ζώνες. Αλλά πρέπει να πούμε ότι τα διάφορα μέσα που εθετούνται για την διαχείριση αυτής ε, αυτού του αλλιεύματος συνεπάγονται πολλές υποχρεώσεις. Όσον αφορά το πού γίνεται η αλληλεία, από πού δραστηριοποιείται κάθε σκάφος, και είναι πληροφορίες που διατίθεται από του εμπορευομένους και επαληθεύονται πληροφορίες από τα κράτη-μέλη σημαία ή από τα άλλα συμβαλόμενα μέρη που έχουν σκάφη που φέρουν τη σημαία τους και που αλλιεύουν σε αυτή την περιοχή. Όσον αφορά το τρίτο ερώτημα, πρέπει να ομολογήσω την άγνοιά μου. Δεν έχω τα αποτελέσματα της συνεδριάσεως που αναφέρατε της χθεσινής συνεδριάς σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ρωμέβα, σημειώνω την ε, πρόσκλησή σας να συναντηθούμε οι δυο μας. Ε, θα καλέσω και τους άλλους και όλους να κάνουν το ίδιο. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο σχόλιο, αν κατάλαβα καλά την Κομισιόν, λέει ότι η απόφαση που πήρε χτε η Κομισιόν σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη της, ε, του ερθρού τόνου στην ΣΥΤΕΣ δεν έχει καταγραφεί σε οποιοδήποτε έγγραφο. Αυτό, θέλει να μου πει η Κομισιόν. Δηλαδή, έχει γνωστή μόνο προφορικά. Πρόεδρος. Φαντάζομαι την απόφαση του κολεγίου των ε, επιτρόπων. Ε, τα πρακτικά δεν ε, δημοσιεύονται, δεν ποτέ πρακτικά δημοσιευμένα από την Κομισιόν, από το κολέγιο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως σας είπα δεν έχω απαντήσει στο ερώτημα, δεν έχω τα αποτελέσματα αυτής της συνεδριάσεως. Είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις και δεν κατέχω αυτά τα στοιχεία. Ωραία, έχω άλλη μια ερώτηση. Κάτι ανεξάρτητο από την έκθεση Ρωμέβα. Υπάρχει το θέμα του κανονισμού 338 που μεταγράφει την κοινοτική ε, την, ε, ε, μεταγράφει σε κοινοτική νομοθεσία τη, τους κανόνες της ΣΥΤΕΣ και είναι πιο περιοριστική, πιο περιοριστικός από ε, την ΣΥΤΕΣ. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την παράκτη αλία που δεν είναι δυνατόν να τύχει εμπορίας εκτός και αν έχει ε, εκτός και αν δοθεί ε, μια εξαίρεση, μια παρέκκληση. Θα ήθελα να δω αν η Κομισιόν θα προβλέψει κάποια τέτοια εξαίρεση ε, γιατί αλλιώς η εραστεχνική αλία που είναι παράκτη αλία δεν είναι δυνατόν να τύχει εμπορίας, να διατεθεί. Έχω, το έχω μελετήσει το θέμα, προσέξτε. η Κομισιόν είναι υπέρ αυτής της παρέκκλησης ή όχι. Γιατί από εκεί θα εξαρτηθεί το κατά πόσον οι εραστέχνες αλληλείς θα μπορέσουν να ε, διαθέσουν το προϊόν τους. Οι παράκτη αλληλείς, εν πάση περιπτώσει. Μπορείτε να μου απαντήσετε, δεν ξέρω τώρα αν εσείς ξέρετε την απάντηση ή αν πρέπει να αναφερθώ, να απευθυνθώ στους υπεύθυνους του περιβάλλοντος. Κυρία Πρόεδρε, πράγματι περί αυτού πρόκειται. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ ο ίδιος σε αυτή την ερώτηση. Το φανταζόμουν. Παρόλο, ε, δεδομένου ότι τη μισή αλία τη χειρίζεται το, ε, το, το, το, το, το χειρίζονται αυτοί του περιβάλλοντος, εγώ γι' αυτό είμαι κατά της ήττες. Εν πάση περιπτώσει, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, για να ανάψουν λίγο τα αίματα. Ήρθα να στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ερώτημα. Το ερώτημα στο οποίο δεν έχω απάντηση. Δηλαδή, αν διέφυγε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Κοινοβούλιο, υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα την ένταξη στο παράρτημα 1 στο ΣΥΤΕΣ υπό προϋπόθεση, δύο προϋποθέσεις που αφορούν δύο τροπολογίες που ψηφίστηκαν μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Η πρω... Ο πρώτος όρος αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του κοινοτικού του ΣΥΤΕΣ, σε συγκεκριμένο πλαίσιο βεβαίως, και όχι με απίστευτους περιορισμούς, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο λοιπόν. Δεν άκουσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τοποθετείται από αυτού. Δεύτερον, δηλαδή το, η συνοδεία οικονομική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς τους ε, πλειοκτήτες και τους ε, ε ναυτικούς που πλήττονται από την ένταξη στο παράδειγμα του ΣΥΤΕΣ. Ε, είμαι ίσως δυσάρεστος έναν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πρέπει να έχετε παρατηρήσει ότι έχει επικυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα λοιπόν οι γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λαμβάνονται υπόψη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά ξεκινάμε άσχημα. Η señora Andrés Barea. Κυρία Άνδρες Βαρέα. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Ενημερώθηκε η, η ΚΑΤ, που είναι ο κατεξοχήν οργανισμός που θα πρέπει να ε, αποφασίζει αν υπάρχουν προβλήματα με τον ερθροτόνο ή όχι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν ανακοινώθηκε στην ε, ΙΚΑΤ ή αν εμείς θεωρούμε ως μοναδικό όργανο διαχείρισης την ΣΥΤΕΣ. Μην ξεχνάτε ότι η ΙΚΑΤ είναι η Διεθνής Οργανισμός Ρύθμισης Αλίας Συνεπώς ε, θα ήθελα να ξέρω ποιε θα είναι οι επιπτώσει που έχει, θα έχει και αν έχει κοινοποιηθεί το κείμενο στην ΕΚΑΤ. Eh, δεν θέλω να δεσμευθεί η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ. Ε, καταλαβαίνω ότι υπάρχει και το θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, αλλά δεν ξέρω, κύριο Μπερζίν, θέλετε να απαντήσετε, έχετε το λόγο. κάνει ανακοινώσεις τακτικές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτά τα αλλιεύματα όπως και άλλα αλλιεύματα. Εδώ υπάρχει ιδιαιτερότης βέβαια διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως γνωρίζετε επιφορτίστηκε με ένα μηχανισμό παρακολούθησης αυτού του αλλιεύματος. Τώρα όσον αφορά το ΣΥΤΕΣ, εάν αυτό το είδος δεν είναι εγγεγραμμένο στο παράρτημα 1, τους ΣΥΤΕΣ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δύναται κατόπιν ιδίας πρωτοβουλίας να κινηθεί. Πρόταση υποβάλλεται, πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα της συνεδριάσεως του αρμόδιου φορέα. Για την ώρα επομίζεται τις ευθύνες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν η κατάσταση όσον αφορά τον ερυθρό τόνο αλλάξει, θα συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της στο νέο πλαίσιο που μπορεί να διαμορφωθεί. Ευχαριστώ. Δεν θέλω να καυγαδίσω μαζί σα. Σας από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ και ε, ξέρω τι σκέφτεστε. Να σα πω όμω το εξή. Το συλλογικό όργανο των, των επιτρόπων, το κολέγιο, πήρε μια απόφαση. Εμένα δεν μου αρέσει, αρέσει άλλου. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πρόταση. Έκανε μια, ε, είναι μια απόφαση να υποβάλει πρόταση. Ε, και μάλιστα οδηγεί σε τροποποίηση κανονισμού του 338. Δεν μπορούμε να προτείνουμε την συμπερίληψη του τόνου στο παράρτημα των απαπειλούμενων ειδών και να μην πούμε ότι θα ε, υποστηρίξουμε την ερασιτεχνική αλία, την παράκτη αλία. Η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της, αυτές που είναι, που υπάρχουν. Συνεπώς, η Κομισιόν θα πρέπει να μας εξηγήσει ποιες θα είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην περίπτωση που θα γίνει δεκτή η πρότασή της. Ανεξάρτητος αν θα εγκριθεί αυτό για τις ΣΥΤΕΣ e ή όχι. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα εγκριθεί η συμπερίληψη του τόνου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Η Κομισιόν όμως υποβάλλοντας την ε, πρότασή της θα πρέπει να λάβει τι ευθύνε τη και να καταστήσει σαφές ποια θα είναι η επίπτωση επί όλων των επιπέδων αν θριαμβεύσει η πρότασή τη, που δεν θα θριαμβεύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι δυνατόν να υποβάλει προτάσει η Κομισιόν ε, που να έχουν σημαντικές επιπτώσει στον τομέα και να μην ξέρουν ποιε θα είναι αυτέ. Απευθύνομαι σε εσά ε, ε, γιατί είσαστε εδώ. Ξέρω ότι θα έπρεπε να είναι η υπεύθυνη του περιβάλλοντο εδώ, όχι εσεί. αλλά εν πάση περιπτώσει. Εμεί έχουμε υποχρέωση να ρωτήσουμε. Γιατί, γιατί μας ρωτάνε και οι, οι, δικοί μας αλλοί. Κυρία Μπαρέα, Αντρέ Μπαρέα, ερώτηση αν έκανε, ε, ε, επέβαλα την ε, ερώτησή μου. η, πρόταση της Κομισιόν υπευλήθη στην ΙΚΑΤ. δεν μου απαντήθηκε αυτή η ερώτηση. Και αν περιμένουν μια, η Κομισιόν περιμένει κάποια απάντηση από την ΙΚΑΤ. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς η Πρόεδρος. Πραγματικό πραγματικός νικητής της συζήτησης ε, στο Κοινοβούλιο είναι η ΚΑΤΕΚ όσον αφορά το θέμα αυτό. Ήταν ηρωνικό αυτό που είπα. Διότι εγώ είχα διαφορετική θέση. Έχασαν οι τροπολογίε μου, περίφθησαν οι τροπολογίε μου. Η ένταξη στο παράρτημα 1 προτάθηκε και φαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το σημείο να λέει καλώ, αλλά σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο διασώζοντας λίγο την τοπική αλληλεία και δίνοντας κάποια χρήματα στους αλληλείς. Και αυτή ήταν η τροπολογία Καντέκ στο Κοινοβούλιο. Εγώ έχω την αντίποση ότι κάνουμε ένα μεγάλο λάθος εκ νέου. Έχω το ξεκάθαρο συνέστημα αυτό. Διότι αν ακολουθήσουμε τη λογική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να επομιστεί αυτό που ψήφισε το Κοινοβούλιο. Εγώ σέβομαι την ψηφοφορία. Θα έπρεπε να πει παράρτημα 1, τελεί και παύλα. Αυτή έπρεπε να είναι η θέση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαφορετικά το Κοινοβούλιο θα πρέπει να οργιστεί, να εξοργιστεί. Έτσι δεν είναι. Θα πρέπει να εκνευριστεί. Διότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να πει όμως παράρτημα ένα σε 12 μήνες και μετά θα παραταθεί θα γίνουν 18 οι μήνες με πόρους που θα πάνε στην αλία που μπαίνουν δηλαδή μπαίνουν από το ένα είδος από τη, από τη σαρδέλα και τα δίνουμε στο, στον τόνο δεν αλλάζει ο πόσο πάει στον τομέα Παίρνουμε από κάπου τα χρήματα και τα δίνουμε αλλού, στον τόνο. Και αυτό είναι δυσκολότατο να γίνει. Διότι εδώ και λίγες μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε το αντίθετο, άλλο πράγμα, ότι δεν υπάρχουν πρόσθετοι πόροι για να διαφυλαχθεί ο τόνος. Ή το ένα το άλλο ισχύει. Καταλαβαίνω ότι η κόσμος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής είναι σε δύσκολη θέση. Διότι ε, βρίσκεται, βλέπει, βομβαρδίστηκε από ανακοινωθέντα τύπου κλπ διάβασα σε κάποια, στον τύπο ότι ναι, σε 12 μήνες θα γίνει αυτό με τοπική διάθεση στο εμπόριο και μετακίνηση των πόρων. Διερωτώ το περιεχόμενο του παρατήματος 2 δεν διαφύλασε, διαφύλασε την τόπια αλία. Ε, εγώ θεωρώ ναι. Η ένταξη στο παράτημα 2 του ΣΥΤΕΣ και δεν προέβλεπε μια φάση κατά την οποία γινόταν έλεγχος του διεθνούς εμπορίου που αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα αυτού που συζητούμε. Πιθανότατα δεν θα έπρεπε να, να συζητούμε την απόφαση του Κοινοβουλίου να μπει ο τόνος στο παράτημα ένα και επιδιώκοντας κι άλλες βελτιώσεις. Εγώ είμαι μέλος επιτροπής Αλίας, αλλά είμαι περιβαλλοντολόγος Είμαι υπέρ του περιβάλλοντος Ποιο είναι το αποτέλεσμα του μπερδέματο αυτού πώς να το πω, με αυτή την απόκληση απόψεων θα, θα φτάσουμε στο ΣΥΤΕΣ, που τα κράτη-μέλη εκεί θα αμελήσουν, θα αγνοήσουν τη θέση της, ε, του Κοινοβουλίου και τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απ' τη μία θα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι και απ' την άλλη τα απομονωμένα κράτη-μέλη, τα ξεχωριστά κράτη-μέλη θα υπερασπίζονται εθνικά συμφέροντα. Εγώ πιστεύω ότι ίσως πάνω σε αυτό, όταν θα συζητήσουμε το θέμα, και θα το αντιμετωπίσουμε συχνά πιστεύω. Ομολογώ δεν εξέτασα προσεκτικά τον κανονισμό. Θα συναγάγω τα συμπεράσματά μου το διαβάσω τον κανονισμό προσεκτικά. Πρέπει να σκεφτούμε παραπάνω πιστεύω. Να βρούμε βελτιώσει και να μην οδηγηθούμε σε αντιπαραθέσει μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι ερμηνεύουν με ακρίβεια τα περιβαλλοντικά θέματα, τα μέλη τη επιτροπή περιβάλλοντο, που έχουν καλά ε, καλές προθέσεις ε, για το περιβάλλον και εμείς εδώ όμως έχουμε ένα επάγγελμα που θέλουμε να διασπιστούμε ε, τη θέση μας. Ε, κυρία Μπιλμπάου, καταρχάς να πω στον κύριο Ρωμέβα ότι θα το συζητήσουμε όπως το κάναμε και με άλλες εκθέσεις μέσω και των τροπολογιών που δεν είχα τη δυνατότητα να προβώ σε ενδελεχή ανάλυση γιατί είχαμε και πιο κατεπήγους εκθέσεις. Λοιπόν, αναλύσουμε αυτή τη σύγχυση ανακοινώσει του τύπου και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει αν θα ενταχθεί το είδο στο παράτημα 1 του σάιτες ή όχι. Τέλο πάντων, να παραδεχτούμε ότι γενικά επικρατεί μια μεγάλη σύγχυση. Αυτό που θα ζητούσα θα ήταν να επικρατήσει διαφάνεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε διαφάνεια. Είναι δική σα ευθύνη να λάβετε απόψει του Κοινοβουλίου αλλά πριν υιοθετηθεί τελική γνωμοδότηση θα πρέπει να κάνετε μια πραγματική διάγνωση των συνεπειών της, των αποφάσεων που λαμβάνονται στην Ευρώπη. Αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να έχει μια σαφή εικόνα σχετικά με τα αλλιεύματα του ερυθρού τόνου ε, στην Ευρώπη την τελευταία πέντα αιτία. Ποιες είναι οι συνέπειες της αποφάσεως να ενταχθεί ο ερυθρός τόνος στο παράρτημα 1 για τις αλληλευτικές κοινότητες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη ιδέα του τι θα κάνει ούτως ώστε να βοηθήσει τους τομείς εκείνους που δεν θα μπορούν να αλλιεύουν ερυθρό τόνο πλέον για τις κοινότητες. Εγώ είμαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλες οι αποφάσεις οι σχετικές με τη μείωση των αλλιευμάτων λαμβάνονται ελεύθερα από όλους, αλλά τομέας για να γίνει πράσινος, να προστατεύει το περιβάλλον, να προστατέψει τα είδη ε, και αυτό έχει σημασία. Αλλά υπάρχει ένας τομέας. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη, να κάνουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Τι αλλιεύματα έχουμε όσον αφορά τον ερυθρότονο στην Ευρώπη, τι ποσότητες. Τι συνέπειε θα έχουν οι αποφάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπής αν πραγματικά πιστεύουν ότι ο ρηθρός τόνο πραγματικά πρέπει να μπει στο παράρτημα ένα του σάιτε. Και τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν τη αυτή περιπτώσει για να βοηθήσει τον τομέα. Ζήτησα και προηγουμένω διαφάνεια και θέλω και εδώ διαφάνεια και σαφεί απαντήσει όσον αφορά αυτά τα ερωτήματα. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή, θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλακερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόγραμμα ήδη το έχουμε συζητήσει για την αλίευση ε, του τόνου. Ελήφθηκε η απόφαση την προηγούμενη εβδομάδα στο Κοινοβούλιο. Δεν ε, συμμετείχαμε όμως εμείς, ε, κυρίως το περιβάλλον είχε λόγο. Δεν νομίζω όμως ότι μας ζητήθηκε καν η γνώμη μας. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι να εκφράζουμε τις απόψεις μας κατόπιν εορτής. Εγώ είμαι από την Ιρλανδία. Εμείς δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο ε, συμφέρον από τον ε, κόκκινο τόνο και ελπίζω αργότερα να μου δώσει απάντηση κομισιόν στο ότι εμείς έχουμε πολύ μικρή ποσόστοση για παραλιεύματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα παραλιεύματα, αν είναι στο ΣΥΤΕ σε εντάξει. Αν υπάρχει, αν αλλιευθεί κόκκινος ερυθρός τόνος, εμείς έχουμε ιδιαίτερα έντονη απόψη για τα απορρίψεις στην Επιτροπή μας και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Και την επόμενη φορά ε, που θα μιλήσουμε για τον ερθρό τόνο, ας δούμε τι θα κάνουμε σε περίπτωση που εμείς παραλιεύσουμε ουσιαστικά κόκκινο τόνο. Εμείς σας λέω και πάλι ότι δεν έχουμε κανένα συμφέρον από τον, από τον τόνο, ε, μόνο στην περίπτωση που ε, υπάρξει κάποια συνέπεια λόγω ε, απορρίψεων. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε τουλάχιστον την ευκαιρία να πούμε μια άποψη για να συμβάλλουμε κι εμείς, γιατί αυτό προς το παρόν δεν έχει συμβεί. Ευχαριστώ. Ωραία. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Ρωμέβα, όλο αυτό είναι αποτέλεσμα ενός ψηφίσματος το οποίο υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλον, ε, Περιβάλλοντος για το site Αυτό γίνεται κάθε χρόνο και ήταν πολύ σημαντικές επιπτώσεις οι φετινές για τον, για τον τομέα της αλίας γιατί συμπεριλήφθη ο ερυθρός τόνος αλλά είναι ένα στάνταρ ε, ψήφισμα που υπάρχει είναι ένα ψήφισμα για την ετήσια ε, συνεδρίαση του site της. Εγώ πάντα το παρακολουθώ γιατί έτσι επισταμένα γιατί ξέρω ότι μπορεί να προκύψουν και θέματα αλληλείας αλλά ίσως να έπρεπε να, καλύψουν, να καλέσουμε συγγνώμη, τους του περιβάλλοντος για να μας πούνε τι ακριβώς συνέβη για με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε κι εμείς να απαντήσουμε Ίσως θα πρέπει να δούμε και τι κάνουν οι άλλες επιτροπές Βέβαια δεν μπορούμε να σταματήσουμε την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος από το να συνάψει αυτό το ε, ψήφισμα, έτσι. Ο κύριος Ρωμέβα έχει το λόγο. Ανέφερα όταν πρωτο, πήρα το λόγο το θέμα αυτό, το πιο σημαντικό είναι το site της. Αλλά για να είμαστε λίγο σοφείς, τα, ε, οι εκθέσεις για τα αλλιεύματα είναι ε, της σημασία, ε, ή μάλλον ο ρόλος που παίζει το site σε αυτές τις εκθέσεις είναι δευτερευούση σημασία. Ε, οι δύο τροπολογίε του site είναι οι 7 και 44. Τι λένε στον κανονισμό που συζητείτε, θα χρειαστεί να γίνουν τροποποιήσεις, προσαρμογές για να συνάδουν όλα αυτά με το site σε περίπτωση που κάτι προκύψει από το site. Οπότε απλώς κοιτάμε λίγο μπροστά Η βάση είναι, ε, η ουσία ουσιαστικά είναι αυτό, είναι η, τα έγγραφα που αφορούν τις, ε, τα αλλιεύματα. Ε, ε, Ωραία. Κλείνουμε αυτό το θέμα. «5 Μαρτίου μέχρι τις 12 το μεσημέρι οι τροπολογίες, 7 και 8 Απριλίου ε, ψηφορία στην Επιτροπή ε, και στην Ολομέλεια του Ιουνίου θα ψηφιστεί οριστικά. Σημείο 8. Όχι 9 λέει πρόεδρος, ε, τη διορθών 8. Σημείο 8. Βιάστηκα λέει πρόεδρος έκθεση σχετικά με την εφαρμογή τη νομοθεσία Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Συντάκτρια η κυρία Λεβίν. Έχετε το λόγο κυρία Λεβίν. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση γιατί εγώ υποχρεώθηκα να κάνω μια έκθεση για μια ε, έκθεση της πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος η οποία ακόμη δεν έχει συνταχθεί. Η Εστέρ Ντελάνζ ακόμη δεν έχει ξεκινήσει ε, με την ε, έκθεση ίδιας πρωτοβουλία για την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Οπότε είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο για να επικεντρωθώ στην βιοπικιλότητα που ε, ένα, σε ένα βαθμό σχετίζεται και με το θαλάσσιο περιβάλλον και με την αλληλεία. Φέτος είναι το έτος του ΟΗΕ για την ε, βιοπικιλότητα, οπότε είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει η έκθεση αυτή, από την Επιτροπή Περιβάλλοντος βέβαια, η εφαρμογή για να επιτευχθούν οι ε, στόχοι για την διατήρηση της βιοποικιλότητας δεν ήταν επιτυχής. Ο στόχος της, ε, της αναστολής ε, της ε, απώλειας βιοποικιλότητας για το 2010 δεν επιτεύχθη. Η απώλεια λοιπόν της βιοποικιλότητας συμβαίνει σε 100 με 1000 φορές περισσότερο από τον συνήθι ρυθμό. Ε, τα τελευταία 50 χρόνια έχουμε χάσει πάρα, πολύ, πάρα πολλά είδη και περίπου 90% της βιομάζας του πλανήτη ζει στους ωκεανούς και πιέζεται συνεχώς. Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καταρχήν έχει ως στόχο να προστατεύσει την ποικιλότητα τους, ε, τους βιοτόπους ε, ε, και να εφαρμόσει την οδηγία για τα πλαίσια για την θαλάσσια πολιτική. Έχουν καθυστερήσει όμως να γίνουν όλα αυτά και αυτό είναι ένας από τους λόγους που δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος. Η αρχική προθεσμία για την εφαρμογή της οδηγίας για τους βιοτόπους ήταν το 1998, πάνω από 10 χρόνια δηλαδή. Και ακόμη δεν την έχουμε επιτύχει αυτή την προθεσμία ακόμη και μετά από 10 χρόνια. Ε, πάνω από 10% των προστατευόμενων ζωνών είναι θαλάσσιες ζώνες στην Ευρώπη και πολλές από αυτές δεν έχουν επαρκή προστασία όταν υπάρχουν μεγάλα, πολλά είδη που ε, ε, τυχάνουν εμπορική εκμετάλλευση όπως το ευρωπαϊκό χέλι και άλλα ε, οι καρχαριοειδοί που δεν αποτελούν μέλος του προγράμματος προστασίας της βιοποικιλότητας παρόλο που υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απειλή και μείωση του πληθυσμού τους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε επίσης ότι η ασυνέπεια μεταξύ των, ε, της βιοποικιλότητας της χερσαίας και της θαλάσσιας ότι δηλαδή η θαλάσσια βιοποικιλότητα δεν ε, την χάνει της ίδιας προστασίας με την χερσαία είναι σημαντικό. Ε, η Κομισιόν έχει καθορίσει κάποιε επιλογέ για ένα νέο στόχο σε μια κοινοποίησή τη που εξεδόθη τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι η Κομισιόν έκανε μια σύνοδο κορυφή στην Αθήνα για τη βιοπικιλότητα με οκτώ συμπεράσματα. Η αλληλεία και οι επιπτώσει τη στη θαλάσσια βιοπικιλότητα αφορούν όλα αυτά τα ε, συμπεράσματα, κυρίω ε, για το αποτύπωμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιοπικιλότητα και την προστασία τη και την ενσωμάτωση όλων αυτών και σε άλλε πολιτικέ. Μείωση τη ε, αλληλευτικής πίεση αναφέρεται πολύ, πολύ συγκεκριμένα ω μία από τι δράσει κλειδιά. Η προστασία τη θαλάσσια βιοπικιλότητα επίση είναι σημαντική για οποιαδήποτε αλληλεία που θα υπάρξει στο μέλλον. Χωρίς ε, οικοσυστήματα υγιή η ε, αλληλεία θα σταματήσει, όχι, αν όχι από του από τους αλλά από του πόρου που θα χαθούν. Πολλά οικοσυστήματα, τα θαλάσσια οικοσυστήματα που είναι υγιή, ε, είναι πιο ανθεκτικά στις πιέσεις, ε, όπως ας πούμε αλλαγές ε, κλιματικές ή ξένα είδη που ενσκύπτουν στους θαλάσσιους οικοτόπους κατακτητικά είδη. Ε, μια που τα κράτη-μέλη έχουν τόσε πολλέ ε, δυσκολίε να εφαρμόσουν ε, την οδηγία για του οικοτόπου και τα πτηνά, ε, πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη υποβολή εκθέσεων για την πρόοδο. Η κοινή αλληλευτική πολιτική πολλέ φορέ καθιστά δύσκολο ή πολλές φορές και αδύνατο να εφαρμόσει κανείς επαρκώς τα μέτρα που χρειάζονται στο, στο Natura 2005 για θαλάσσιους τομείς. Αυτή λοιπόν είναι η φάση που χρειαζόμαστε περιορισμούς στην αλληλεία έτσι ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε την οδηγία για τους οικοτόπους. Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα στη δική μου γνωμοδότηση. Η κοινή, αγρο... η κοινή αλληλευτική πολιτική δεν θα πρέπει να δυσκολεύει, θα πρέπει να διευκολύνει τις υποχρεώσεις για την ε, προστασία των ε, θαλασσιών περιοχών δεν έχει υπάρξει επιτυχία λοιπόν στην μείωση των, της υπεραλίευσης των γόνων, των θαλασσίων φυλαστικών, των χελωνών και των θαλασσίων πουλιών. Και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει δράση κλειδί στην πολιτική μας και πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας ακόμη περισσότερο. Η γνωμοδότησή μου είναι αρκετά σύντομη. Μια σελίδα είναι, όλοι και όλοι. Ο κύριος Αρσένης ε, ξέρει ακριβώς τι είναι. Και βεβαίως, εάν έχετε τροπολογίες, ευχαρίστως να τις λάβω για να προσθέσουμε και άλλες ε, σημαντικές πληροφορίες στη γνωμοδότηση. Τέλος, να πω ότι τα σχολεία της κυρίας Μπιλβάου για το ότι είναι δωρεάν να είναι κανείς περιβαλλοντολόγος ε, εγώ δεν συμφωνώ. Δεν, η φύση τουλάχιστον δεν είναι δωρεάν. Και αν μπορούμε να έχουμε και κάποια οικονομική, ένα οικονομικό αντιστάθμισμα προς τους πολίτες μας που και τώρα ζουν και στο μέλλον θα ζουν στη φύση που ίσως να μην μπορούμε βέβαια να το μετρήσουμε ίσως να το έχουν προσπαθήσει κάποιοι οικονομολόγοι του ΟΗΕ βέβαια αλλά μάλλον σε ό,τι αφορά το πόσιμο νερό, τον καθαρό αέρα ε, και τα αλλιεύματα που ούτως ή άλλως είναι τρόφιμα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το συγκρίνουμε με οποιοδήποτε ΑΕΠ. Και να συγχαρώ τον κύριο Αρσένη για την γνωμοδότησή του για την κλιματική αλλαγή που τονίζει ακριβώς αυτό που είναι πολύ σημαντικό, ότι τα υγιή οικοσυστήματα στους ε, ωκεανούς μας έχουν μεγάλο δυναμικό απορρόφησης διοξιδίου του άνθρακα που μπορεί να αναστείλει την κλιματική αλλαγή. Και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σαρσένης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ε, πραγματικά τα... θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ με την σειρά μου την κυρία Λοβάν για την εξαιρετική δουλειά της ε, υπό πραγματικά αντίξωες συνθήκες ε, από τη στιγμή που δεν υπάρχει η βασική έκθεση. Ε, πραγματικά έχει, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βιοπικιλότητα έχει αποτύχει παταγωδός. Ε, είχαμε ως στόχο μέχρι το 2010 στην ουσία να σταματήσουμε, ε, να σταματήσουμε την απώλεια βιοπικιλότητας και χάνουμε, συνεχίζουμε να χάνουμε ήδη με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Συμφωνώ με όλα τα σημεία της έκθεσης της κυρίας Λοβάν. Θα ήθελα να προσθέσω μερικές ε, ιδέες. Ένα βασικό σημείο που νομίζω θα άξιζε να είναι στην έκθεση είναι η οικοσυστημική προσέγγιση ως βασική αρχή της πολιτικής για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και για την αποκατάστασή της. Ε, θα νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αναφορές για την ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών και για το, μιας και ο σεβασμός της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων είναι πάρα πολύ βασικός. Ε, είναι σημαντικό πάντοτε να, να στοχεύουμε σε ένα, στην κατάρτιση άμεσα, το γρηγότερο δυνατό και υλοποίηση ενός σχεδίου αποκατάστασης κιόλας βιοποικιλότητας. Ε, όπως είπε η κυρία Λοβάν, οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές είναι πολύ σημαντικές, πρέπει να ολοκληρωθούν. Χρειαζόμαστε ένα συνολικό και συνεκτικό δίκτυο θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών πολύ βασική, ε, κατά τη γνώμη είναι η αρχή της ισοτιμίας, ε, η οποία χρειάζεται να εφαρμοστεί ε, στα πλαίσια που συζητάμε. Διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης έχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά μέτρα χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας, αλλά και η αποκατάστασή της σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, μπορεί να ωφελούμαστε όλοι από τη βιοπικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές και θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τρόπους ε, ανταμοιβή των περιοχών, που, των ε, περιοχών της Ευρώπης, των κατοίκων των περιοχών της Ευρώπης που έχουν ε, προστατεύσει τη βιοπικιλότητά τους και χάρη στις υπηρεσίες που προσφέρουν αυτοί ε, είμαστε και εμείς σε θέση να απολαμβάνουμε πάρα πολλά αγαθά που όπως είπε η κυρία Λοβάν κοστίζουν πάρα πολύ αν θέλαμε να τα παράξουμε μόνοι μας. Επίσης, θα πρέπει πάντοτε να κοιτάμε ότι όταν λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αυτά δεν θα έχουν αρνητικές συνέπειες στη βιοπικιλότητα. Η προστασία της βιοπικιλότητας είναι προϋπόθεση για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Χρειαζόμαστε ε, την ανάπτυξη επίσης στρατηγικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της εισβολής και εξάπλωσης ξένων ειδών. Τέλος, στα πλαίσια και των συζητήσεων που είχαμε για άλλα θέματα και στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο, πραγματικά χρειαζόμαστε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τα αντισταθμιστικά ωφέλη ε, και τη χρηματοδότηση των παραγωγικών ομάδων που θα, που θα χθιχθούν στην ουσία, θα, δεχθούν, θα έχουν αρνητικές συνέπειες από τη λήψη των ε, νέων μέτρων για την προστασία της βιοποικιλότητας που αν και είναι μια, αυτόνομη, μια, αυτο, μια αυτονόητη αρχή, ε, μόλις τώρα αρχίζουμε να την εξετάζουμε σοβαρά. Κυρία Φράγα, πριν δώσω το λόγο σε άλλους ευρωβουλευτές, να καλωσορίσω μια ομάδα Γερμανών φοιτητών από το Μόναχο. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρον το θέμα μας παρόλο ότι ε, η Βαβαρία δεν είναι και η πιο συνδεδεμένη <laughs> με τον κόσμο της ε, αλληλείας περιοχή της Γερμανίας, ούτε η Γερμανία στο σύνολό της βέβαια. πάση περιπτώσει η συζήτηση είναι αρκετά ζωντανή ε, και έχουμε και μια ποικιλία θεμάτων. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι οι φοιτητέ να έρχονται στην Επιτροπή μας, μικρή αλλά δραστήρια. Κανείς άλλος δεν έχει ζητήσει το λόγο. Να κάνω τότε εγώ κάποια σχόλια. Πρώτον, σημείο 9. Αυτό που είπα και στον κύριο Ρωμέβα. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε συζήτηση για το θέμα αυτό, αλλά αυτό που είπα και στον κύριο Ρωμέβα ισχύει και στη, για τη δική σας νομοδότηση. Δεν συμφωνώ με το 9. Δεύτερον, θα μπορούσαμε να τονίσουμε λίγο περισσότερο το εξής κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την προάσπιση της βιοπικιλότητας στο δικό μας τομέα, που είναι το, η οικοσυστημική προσέγγιση. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση θα μας βοηθήσει στην διατήρηση της βιοπικιλότητας. μέσω αυτής της προσέγγισης θα δημιουργήσει επιστημονική έρευνας και άλλες μέσω των οποίων θα προασπίσουμε καλύτερα την βιοποικιλότητα. Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η σύνδεση στον ε, κλάδο της αλίας. Εκ μέρους της Κομισιόν ο λόγος στον κύριο Παπούλια. Ολαθάβαλ. Α, Ολαθάβαλ, όχι Παπούλιας, Ολαθάβαλ. Αλλάξαμε και φίλο και ε, εθνικότητα και απ' όλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, δύο στην τιμή του ενό, γιατί ο κ. παπούλια θα μπορούσε να σχολιάσει το θέμα τη εφαρμογή του Natura 2000. Καλωσορίζουμε την, το σχέδιο γνωμοδότησης Κυριά Λεβίν. Καταλαβαίνουμε πολύ πόσο δύσκολο είναι να γράψει κανεί κάτι χωρί να έχει την έκθεση τη κυρία Ντελάγκε. Είναι και επίκαιρη στιγμή γιατί το Συμβούλιο συζητάει τις επιλογές για το στόχο του 2020 και, και την προθεσμία του 2050. Συνεπώ είναι πολύ σημαντικό αυτές οι νομοθεσίες του Κοινοβουλίου να συμπληρώσουν τις ε, συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή βεβιασμένα σε μεγάλο βαθμό στο Συμβούλιο γιατί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου θα υιοθετηθούν στις 15 Μαρτίου για αυτό το θέμα. Συμφωνούμε με τα περισσότερα από όσα είπε η κυρία Λεβίν και αναφέρει στην έκθεσή της. Άλλωστε τα έχουμε υπογραμμίσει και εμείς ε, στην ανακοίνωση Επιτροπής τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα πετύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει για το 2010. Δεν καταφέραμε να ανασχέσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απώλεια βιοπικιλότητα συνεχίζεται, απώλεια οικοσυστημάτων ε, συνεχίζεται και το εκτιμόμενο κόστος είναι 50 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την απώλεια αυτών των οικοσυστημάτων. Οπότε και από οικονομική ε, πλευρά, αν το δούμε μόνο, είναι πολύ ανήσυχο το πανόραμα. Ανησυχητικό το πανόραμα. Για όσου δεν το γνωρίζουν από εσά, να σα πω ότι υπάρχει μια τεράστια πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα. Είναι μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία οικονομολόγων που χρηματοδοτείται από την Κομισιόν, την γερμανική κυβέρνηση και την βρετανική κυβέρνηση και έχει ω στόχο να αξιολογήσει την οικονομική σημασία των, ε, της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Στόχος ε, είναι η βιοπικιλότητα ε, να ενταχθεί στις πιο παραδοσιακές οικονομικές συζητήσεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα της εφαρμογής, η Κομισιόν έχει πει ότι οι οδηγίες ε, πτηνών ε, οικοσυστημάτων και ύδατο ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως ως τμήμα οποιοδήποτε στόχου βάλουμε στον εαυτό μα για το μέλλον. Οποιαδήποτε ε, πλημελής εφαρμογής τους θα πρέπει να μας υποδειχθεί. Και γι' αυτό το λόγο θα δώσω το λόγο στον κύριο Παπούλια που μπορεί να καλύψει και το θέμα των προστατευόμενων θαλάσσιων ζώνων. Ευχαριστώ. Και εγώ καλωσορίζω αυτή, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης που ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις δικές μας τρέχουσες πρωτοβουλίες, ε, ε, συγγνώμη. Θα ήθελα να εστιαστώ λίγο στα, ε, στο Natura 2000. Η Κομισιόν ανησυχεί ιδιαίτερω για σημαντικές καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τον επαρκή καθορισμό ζωνών Natura 2000, ε, θαλάσσιων ζωνών στο πλαίσιο του Natura 2000. Ιδιαίτερο στην ανοιχτή θάλασσα, ε, εκτός δηλαδή των ε, εγχώριων υδάτων. Στις πρώτες, στα πρώτα χρόνια εφαρμογής των οδηγιών για τα πτηνά και τα και τα οικοσυστήματα ε, ε, εστιαστήκαμε στις χερσαίες ζώνες γιατί είχαμε περισσότερη γνώση αλλά τα τελευταία χρόνια ε, έχει πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί η εργασία του χερσαίου τμήματος του Natura 2000 και γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν έχει ως προτεραιότητα την επέκταση του Natura 2000 και των δράσεων στις θαλάσσιες ζώνες. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο το δίκτυο Natura 2000. Χαίρομαι που μπορώ να πω ότι ολοκληρώνουμε αυτή την εποχή την ε, κοινοτική ε, διαδικασία ε, για την επιλογή βιογραφικών σεμιναρίων. Φέτος θα έχουμε καλύψει πλέον όλες τις ευρωπαϊκές θάλασσες με αυτή την επιστημονική, σφαιρική επιστημονική αξιολόγηση. Αυτή η διαδικασία θα μας παράσχει βάσιμα επιστημονικά στοιχεία για να προσδιορίσουμε τα κενά που έχουν αφήσει μέχρι τώρα οι προτάσεις των κρατών μελών. Η Κομισιόν θα πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να ενθαρρύνει τα κρατη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για την συμπλήρωση των θαλασσιών ζωνών. Το άλλο κομμάτι αφορά την διαχείριση των θαλασσιών ζωνών Γνωρίζουμε τις ε, προκλήσεις του που αντιμετωπίζουν αυτές οι ζώνες, ε, δέχονται πιέσεις ε, παντιοτρόπως. εξαιτία πολλών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται όλο και περισσότερο στις θαλάσσιες ζώνες, ιδιαίτερο στην Αλία. Η Κομισιόν έχει εκδώσει ε, τις γραμμές το 2006 για το θέμα της διαχείρισης ε, των θαλασσιών ζωνών. Η πρόθεσή μας είναι να δώσουμε στα κράτη-μέλη τις δυνατότητες και την ενθάρρυνση να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ε, προκειμένου να τροποποιηθούν οι ισχύουσε πρακτικές, ε, να επιβληθούν απαγορεύσει ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο που αφορά την αλία σε ζώνες που προστατεύονται. Επίσης ε, ετοιμάσαμε και κατευθυντήριες ε, γραμμές για να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη στην προετοιμασία μέτρων που λαμβάνουν στην Αλία στο πλαίσιο της κοινή αλληλευτικής πολιτικής ε, για να διευκολύνουν δηλαδή, τα κράτη-μέλη ε, σε, όλο αυτό το, σε όλη τους αυτή την προσπάθεια. Υπό το φως των εμπειριών, ε, μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί, σκοπεύουμε να βελτιώσουμε μάλιστα στο μέλλον αυτές τις κατευθύνσεις γραμμές. Να προσθέσω τέλος ότι σε σχέση με άλλες θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες, που προβλέπονται από την οδηγία της ε, ε, θαλάσσιας στρατηγικής. Στόχος μας είναι να συντονίσουμε ε, τις προσπάθειές μας στο πλαίσιο του Νατρίου 2000 μαζί με τις προσπάθειες ε, που κάνουν άλλες συμβάσεις, η ΟΣΠΑΡ, η Σύμβαση της Βαρκελόνης, για άλλου τύπου και άλλες προστατευμένες ε, περιοχές. Θα συνεργαστούμε με αυτούς τους διεθνείς φορείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να τελειώσουμε. Ε, Κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Η ιδέα αυτή για το ότι χρειαζόμαστε σχέδια για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις παράκτητες περιοχές είναι καλή. Βέβαια δεν θα, μπορούσαμε να μιλάμε για πάντα για τα οικοσυστήματα. Νομίζω όμως ότι όντως είναι σωστό αυτό που λέτε ότι πρέπει να τα τονίσουμε ακόμη περισσότερο. Χαίρομαι που η Κομισιόν και το Συμβούλιο θεωρούν ότι βαδίζω προς τη σωστή κατεύθυνση. Οπότε το μόνο που μου μένει εμένα είναι να συνεχίσω τη δουλειά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Λουβίν. 3 Μαρτίου η υποβολή ε, τροπολογιών και 7 και 8 θα γίνει η ψηφοφορία. Πάμε στην επόμενη. Στο επόμενο θέμα, σημείο 9. Χρήση ξένων και απόντων σε τοπικό επίπεδο ειδών στην υδατοκαλλιέργεια. Ο κύριος Ζωάου Φερέιρα είναι ο εισηγητής. Στην τελευταία συνεδρίαση ακούσαμε την πρόταση της Κομισιόν. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή για να μας πει την απόψή του και μετά θα το συζητήσουμε. Eh, um Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για την διατήρηση της βιοπικιλότητας μόλις και το θέμα αυτό συνδέεται με το δικό μου. Όλοι γνωρίζουν πως ε, τα ξένα είδη είναι ένας από τους ε, παράγοντες της ε, απώλειας βιοποικιλότητας. Καταστρέφουν τους οικοτόπους. Υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι απώλειας βιοποικιλότητας. Ένας είναι τα ξένα είδη και ένας είναι άλλοι λόγοι που καταστρέφουν τα οικοσυστήματα. Αυτό που προτείνει τώρα η Κομισιόν είναι η τροποποίηση του κανονισμού 708 κάθετος 2007 θα επαναπροσδιορίσουν τι σημαίνει κλειστό κύκλωμα στην ε, υδατοκαλλιέργεια για να αποφευχθεί η ε, εισβολή ξένων και απόντων ειδών. Ο στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υδατοκαλλιέργεια και να διευκολυνθούν όσοι δρούν στον τομέα αυτό. Και να γίνει αυτό με τρόπο που να μην είναι επαχθής. Η κείμενη νομοθεσία επιτρέπει εξαιρέσεις για την ε, αποκτησία αδειών στην ιδιωτοκαλλιεργία για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται σε κλειστό κύκλωμα. Αυτό επί τη βάση νέων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων και πληροφοριών Υπάρχει και το πρόγραμμα IMPAS, το οποίο χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του έκτου προγράμματος πλαισίου και περιέλαβε πολλούς ε, οργανισμούς και ως τμήμα του ε, προγράμματος αυτού υπάρχει νέος ορισμός των κανόνων που εφαρμόζονται για την ιδιωτοκαλλιέργεια κλειστού κυκλώματος και τις εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες για την βιοασφάλεια τηρούνται. Είναι πιο αυστηροί και πιο λεπτομερείς. Ε, έτσι αποφεύγεται οποιαδήποτε αμφιβολία υπάρχει, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το είδος αυτών των εγκαταστάσεων και την, ε, της εδωτοκαλλιέργειας ε, την οποία, η οποία εκτιλήσεται μέσα από αυτές τις εγκαταστάσεις. Οπότε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύμφωνα με το πρόγραμμα IMPAS, ο ορισμός του κλειστού κυκλώματος και, της και των σχετικών ε, εγκαταστάσεων θα μειώσει τον συσχετισμό με τα ξένα και απόντα είδη και θα τα φέρει σε ένα ε, επιτρεπτό επίπεδο. Αξιολόγηση κινδύνου έγινε επί τη βάση μιας τεχνικής αξιολόγησης και το κατά πόσο θα γίνει αποδεκτό αυτό ή όχι, το επίπεδο κινδύνου δηλαδή, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Πέρα από αυτό, αυτό που λέει η Κομισιόν είναι ότι το πρόγραμμα IMPAS επιτρέπει μείωση κινδύνου ώστε να είναι πολύ χαμηλότερη από αυτούς που έχουμε τώρα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν εδώ τα πράγματα. Η Κομισιόν αναγνωρίζει το προγραμμα ιμπας επιτρεπει μειωση κινδυνου ωστε να ειναι πολυ χαμηλοτερη απο αυτους που εχουμε τωρα υπαρχουν πολλοι παραγοντες που επηρεαζουν εδω τα πραγματα η κομισιον αναγνωριζει το γεγονος πως ε, για παράδειγμα οι μεταφορές και η συμμόρφωση με τις διαδικασίες που καλύπτουν τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η λειτουργία τους ε, λοιπόν και η δομή τους και οι κανόνες που τους διέπουν ε, είναι πολύ αυστηρά τα πρωτόκολλα που ασχίουν για τις ε, συγκεκριμένες υδατοκαλλιέργειες αλλά η μεταφορά αυτών των προϊόντων επίσης καλύπτεται και αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη. Θα ήθελα να ακούσω επίσης την γνώμη της Κομισιόν σε σχέση με μια κρίσιμη πτυχή που έχει σχέση με την εξακρίβωση της συμβατότητας αυτών των ε, μάλλον της εφαρμογής αυτών των κανόνων σε μελλοντικές εγκαταστάσεις που θα ανοίξουν στο μέλλον. Ποιος δηλαδή ε, θα εξακριβώνει την τήρηση αυτών των κανόνων σε νέες εγκαταστάσεις. Ποιος θα κάνει δηλαδή το monitoring, την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών των κανόνων. Να πω επίσης ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη μια σειρά γνωμοδοτήσεων όπως η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ δεδομένου το άρθρο 42 της Συνθήκης Λισαβόνας προβλέπει υποχρεωτικά την έκδοσή της και μια η οποία γνωμοδότηση ΟΚΕ ε, θέτει μια σειρά θεμάτων που κατά την άποψή μου είναι πολύ σωστά. Θα πρέπει λοιπόν να λυθεί υπόψη η γνωμοδότηση τη ΕΟΚΕ, καθώς επίση και μια σειρά άλλων γνωμοδοτήσεων που έχουν εκδώσει στο παρελθόν τεχνική και μυρογνώμονα στο τομέα. Ευχαριστώ. Κύριος με την επιφύλαξη των ε, απόψεων για τη βιοπικιλότητα και των ε, θέσεων της ε, εισηγήτριας, ο στόχος είναι οι κλειστές ηχθειοκαλλιέργειες να εξαιρεθούν. Πρόκειται για μια καινούρια διάταξη για αυτού του τύπου της. Ε, εγκαταστάσεις. Εμείς είμαστε υπέρ οποιαδήποτε μείωση γραφειοκρατίας. Ε, νομίζω ότι η διάταξη αυτή δίνει ε, μεγαλύτερη ελαστικότητα βέβαια συνοδευόμενη από τις επαρκείς εγγυήσεις περιβαλλοντικής προστασίας. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμος αυτός ο κατάλογος των κλειστών χθιοκαλλιεργιών οτιδήποτε μειώνει τη γραφειοκρατία, μειώνει τα ε, κόστη τα σχετικά με την ε, κόρηση αδειών που συνοδεύεται όμως από επαρκείς περιβαλλοντικές διατάξεις προστασίας ε, μας φαίνεται θετικό. Ευχαριστώ. Eh, κύριε Λεβίν. Σας ευχαριστώ. Διερωτώ για το σημείο αυτό της μειώσεως της γραφειοκρατίας και της μειώσεως του κόστους για τον τομέα. Κύριε Φέιρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχετε πληροφορίες για το κόστος. Ποιο είναι το τρέχον κόστος για την αδειοδότηση. Πόσο σημαντικό είναι το ποσό, πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Πρέπει να ζητήσει κανείς άδεια μία φορά κάθε περίοδο, κάθε εποχή ή άπαξ απαντός άμα ξεκινά κανείς τη δραστηριότητά του. Και διαρωτώ με κατά πόσο περικόπτεται κατά πολύ γραφειοκρατία αν πρόκειται περί μιας και μοναδικής αδείας. Το ξεκινά κανείς τη δραστηριότητά του. Έχω και πρόβλημα όσον αφορά τους ορισμούς για τις ασφαλείς εγκαταστάσεις. Θα πρέπει να καθορίζονται οι κανόνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής ή τα κρατημέλη θα μπορούν να επηρεάσουν το, τον καθορισμό του κλειστού συστήματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριος Σκουέφ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι η Επιτροπή σας συνόψισε τέλεια την όλη προβληματική. Δηλαδή θέλουμε να προσμετρήσουμε το κόστος ε, Διαχείριση ενός συστήματος που είναι πολύ επαχθές διοικητικά, η μετακίνηση αυτών των ειδών που επηρεάζει την αδειοδότηση είναι κάτι πολύ επαχθές. Χρειάζεται μια επιτροπή αξιολογήσεως του κινδύνου και μετά που θα κάνει την αξιολόγηση να δώσει την άδεια. Το θέμα που ετέθη ευθύ εξ αρχή όταν συζητήσαμε τον κανονισμό ήταν το εξή. Να απαλλάξουμε αυτά τα κλειστά συστήματα όσον αφορά τον κίνδυνο διαφυγής υλικού ε, γενετικού από ε, την ηχθειοτροφία. Να προβλέπετε ένας ορισμός ο οποίος θα είναι συγκεκριμένος για τα κλειστά συστήματα ώστε να περιορίζεται ο διοικητικός κίνδυνος όσον αφορά τη σωστή αξιολόγηση του κίνδυνου. οδηγηστήκαμε στο αδιέξοδο όσον αφορά τον ορισμό του κλειστού συστήματος. Χρειάζεται μεγάλη ακρίβεια, πολλή τεκμηρίωση. Κατά την άποψή μας, κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην τροποποίηση του κανονισμού για την εισαγωγή τομή ε, ντόπιων ειδών ε, μπορούμε να προβλέψουμε κανόνες ε, μέσω του, των εσωτερικών ορισμών. Ξέρουμε ποιο είναι το διοικητικό κόστος όσον αφορά την έκδοση αδείας. Όχι πραγματικά. Αυτό συνεπάγεται εμπλέκει της υπηρεσίες της ήδη υπάρχουσες. Δύσκολο να εκτιμηθεί το κόστος αλλά κατά ομόφωνη άποψη θεωρούν ότι το κόστος είναι μεγάλο τα κράτη-μέλη και πρέπει να κάνουμε οικονομίες εκεί που δεν υπάρχει πλέον κάποιος κίνδυνος. Θα ήθελα να πω επίσης ότι είμαστε στη διάθεση του κυρίου Φερέρα, του συγγητού, για επαφέ για να δώσουν περισσότερε πληροφορίε που μπορούν να του είναι χρήσιμε για να συντάξει την έκθεσή του. Αυτά και ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριο Φερέρα για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύριος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και την Κομισιόν για τα σχόλιά τους. Αντιλαμβάνομαι τα θέματα τα οποία ε, έθεσε η κυρία Λέβιν. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα. Το 20% των εξωτικών ειδών που εισάγονται σε εσωτερικά ύδατα προέρχονται από υδατοκαλλιεργίες. Συνεπώς το θέμα είναι ευαίσθητο. Ε, ας μην κάνουμε όμως ε, τα κριτήρια ε, πάρα πολύ αυστηρά. Μπορεί δηλαδή να μειώσουμε τον κίνδυνο της διαφυγής εξωτικών ειδών αλλά να μην είμαστε υπερβολικά αυστηροί διότι θα πρέπει να αποφύγουμε οποιοδήποτε περιτόγραφιο κρατικό άχθος. Ίσως χρειάζεται όμως να συμπεριλάβουμε, να προσθέσουμε κάποιες διατάξεις ό,τι αφορά την παρακολούθηση της λειτουργίας και της αδειοδότησης αυτών των εγκαταστάσεων. Αυτό ίσως πράγματι είναι απαραίτητο, ναι, πολύ κρίσιμο. Να εγγυηθούμε δηλαδή ότι οι εγκαταστάσεις θα τηρούν τους κανόνες που υφίστανται. Θα ήθελα να κάνω και μια παρατήρηση, μια πρόσθετη παρατήρηση για την ανάγκη επίγουσα πιεστική ανάγκη στην οποία επιμένουν ειδικοί και διάφορα Ινστιτούτα ερευνητικά κλπ. Μου ελέγχθη ότι υπάρχει έλλειψη υποστήριξης επιστημονικής έρευνας για αυτόχθονα είδη θεοκαλλιέργειας γιατί η εισαγωγή στην ε, ηχθειοκαλλιέργεια εξωτικών ειδών που είναι απόντα από το τοπικό επίπεδο χρειάζεται ε, συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Πολλά κέντρα ερευνητικά κλπ. ακολουθούν αυτή την οδό. Και η αλήθεια είναι ότι η εισαγωγή τέτοιων ειδών ε, δημιουργεί εξασφαλίζει μεγαλύτερη ποικιλία διατροφική, καινούργια προϊόντα στην αγορά κλπ. Αλλά αυτά τα επιστημονικά κέντρα πέραν των πρωτοκόλων που δεν υπάρχουν και προσπαθούν να αναπτύξουν για μια αυτόχθονα είδη, θέλουν να αναπτύξουν πρωτόκολλα και για αυτόχθονα είδη, αλλά έχουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. Χρειάζεται λοιπόν να υποστηρίξουμε και την επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτό. Μου το ανέφεραν πολλά επιστημονικά ιδρύματα. Το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας δύσκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου ε, ποσά και κονδύλια να διοχετευτούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Φερέιρα. Θα μας υποβάλλετε την έκθεσή σας. Θα τη δούμε στην επόμενη συνεδρίασή μας. Κλείνουμε και το 9. Περνάμε στο σημείο 10 της ημερησίας διάταξης, τελευταίο για το πρωί ενημέρωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού 1967-2006 σχετικά με τις τεχνικές διαχείρισης και διατήρησης στην Μεσόγειο. Ε, αυτό έχει σχέση με μια επιστολή που έστειλε η Κοζέκα στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου εξέφραζε ανησυχία για τρία θέματα το μέγεθος του ματιού, τις ελάχιστες ε, αποστάσεις που καθορίζει ο κανονισμός και τρίτον το μέγεθος του του Μπόρατς δεν κατάλαβε ο διερμηνέας τι εννοούσε η πρόεδρος. Ε, θα ήθελα η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή να μας ενημερώσει σε σχέση με αυτές τις ανησυχίες της ΚΟΖΕΚΑ ε, οι οποίες ε, ανησυχίες σχετίζονται με όλη τη Μεσόγειο. Ο κύριος Λάμπελ Μάιερ έχει το λόγο. Eh, euh, Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε για να συνημερώσουμε επί του κανονισμού που για μας είναι σημαντικότατος και για την Αλία και τους Αλίες της Μεσογείου και είναι και μια ευκαιρία να μιλήσουμε γενικά για την Αλία στη Μεσόγειο. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείχνετε για το θέμα κάτι που συμμεριζόμαστε απόλυτα, ξέρετε σίγουρα και θα θυμόσαστε ότι η νέα Επίτροπος, όπως και η προκάτοχή της, προσδίδει μεγάλη σημασία στην ε, αλληλεία στη Μεσόγειο και ενδιαφέρεται όλους ιδιαίτερα το θέμα. Αληθεύει ότι η Μεσόγειος όσον αφορά την αλληλεία δεν είναι στο προσκήνιο, δεν εμφανίζεται πολύ συχνά στο προσκήνιο, διότι στη Μεσόγειο δεν έχουμε το περίφημο ετήσιο ραντεβού για τον καθορισμό ποσοτήτων, ποιοτικών ε, ποσοτήτων, ποσοστώσεων ποσοτικών, τα περίφημα τάκ, αλλά ακολουθούμε διαφορετική προσέγγιση στη Μεσόγειο και έτσι πηγαίνω στον ίδιο τον κανονισμό. Ίσως δεν απόλυτα σωστό να αποκαλείται κανονισμός τεχνικών μέτρων, διότι είναι και ένας κανονισμός τεχνικών μέτρων, αλλά και πολλά περισσότερα. Στην πραγματικότητα είναι ένας κανονισμός ο οποίος μπορεί να καυχηθεί ότι είναι ο πρώτος ε, κανονισμός που ακολουθεί ολοκληρωμένη προσέγγιση οικοσυστημική. Ε, οικοσυστημική. Λοιπόν, εμπεριέχει καταρχάς ε, διατάξεις οι οποίες έχουν σαν στόχο την προστασία των ειδών και των βιοτόπων και άλλων κάνει άμεση διασύνδεση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και ανταποκρίνεται στην υποχρέωση να συμπεριληφθούν οι περιβαλλοντικές πτυχές σε όλες τις πολιτικές. Και δεύτερον, αυτός ο κανονισμός στοχεύει σε μια νέα προσέγγιση διαχείρισης κάτι που συζητήσαμε πρόσφατα στους τελευταίους μήνες, διότι τονίζει ο κανονισμός μια προσέγγιση εκ των κάτω προς τα πάνω, δηλαδή η περίφημη προσέγγιση bottom-up και δίνει πρωταρχικό ρόλο στην τοπική αυτοδίκηση. Και στα κράτη-μέλη βεβαίως, που πρέπει να δώσουν εθνικά σχέδια διαχείρισης όσον αφορά την αλληλεία τους αλλά και προτάσεις που θα καθορίζουν προστατευμένες ζώνες στα ύδατά τους και πέραν αυτών. Είναι μια προσέγγιση περιφερειακή που προσαρμόζεται πολύ καλά ή θα μπορούσε να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες στις διάφορες και όσον αφορά και τη μερίθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής πρόκειται περί πρώτης εφαρμογής της νέας προσεγγίσεως που αποφασίστηκε αλλά τρία χρόνια μετά από την θέση σε ισχύ του κανονισμού η εφαρμογή του δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική, νομοθετικός και πρακτικός. Τα διαχειριστικά σχέδια, όλα τα κράτη-μέλη πράγματι υπέβαλαν τέτοια σχέδια ή καμιά φορά αυτό που αποκαλούν σχέδιο, αλλά αυτά τα σχέδια δεν ανταποκρίνονται όλα δυστυχώς στα αναγκαία κριτήρια, δηλαδή η σωστή επιστημονική βάση, καλή περιγραφή της αλίας, και των ενδειγμένων μέτρων και για τον καθαρισμό των προστατευμένων ζωνών και εκεί λάβαμε κάποιες προτάσεις αλλά η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική όσον αφορά ε, το δίχτυ, τον τετραγωνισμό, τον διαχωρισμό. Ε, το 2009 είδαμε ότι υπάρχει κάποια εφαρμογή ήδη ο ίδιος ο κανονισμός εμπεριέχει και κάποια παρέκκληση για το μάτι των δικτύων, το τετράγωνο. Ε, μέχρι το Μάιο 2010 πρέπει να εφαρμοστούν τα μέτρα. Ε, δεν εφαρμόζεται υποχρεωτικά ακόμα, όλος ο κόσμος θα ακολουθεί, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές παρεκκλήσεις και θεωρήθηκε ότι πρέπει να υπάρξει μεταβατική περίοδος για να εφαρμοστεί ο νέος κανόνας για τα δίκτυα. Τώρα όσον αφορά το μάτι των δικτύων το τετράγωνο ή το ρομβοειδές τα κράτη-μέλη μας διαβεβαιώνουν ότι είναι καθοδόν εφαρμόγη. Λοιπόν, μας εξέπλησε κάπως η προσέγγιση του ΚΟΣΕΚΑ, όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, και δεν συμφωνούμε καθόλου με την ανάλυση που γίνεται εκεί. Επιτρέψτε μου να προσθέσω ένα τελευταίο σχόλιο. Η Μεσόγειος ε, έχει μεγάλη ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα κοινοτικά ύδατα. Όπως γνωρίζετε δεν υπάρχουν κοινοτικά ύδατα, υπάρχουν ε, κρατικά ύδατα και όχι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες. Γι' αυτό λοιπόν ακολουθούμε μία προσέγγιση διτή. Από τη μία πλευρά με τον κανονισμό που έχουμε τον κανονισμό για τη Μεσόγειο, για τον κοινοτικό κανονισμό, αλλά ε, και στα ύδατα η ΚΑΤ σε άλλα ύδατα, σε ΖΕΠΕΜ που αναφέρατε ήδη επανειλημμένα. Έχουμε πρόταση να εφαρμοστούν τα σχετικά μέτρα και ήδη τα καταφέραμε να υιοθετήσουμε κάποια σύσταση στη ΣΕΖΕΠΕΜ ε, που έχουμε το κοινοτικό κεκτημένο των δικτύων των 48 μέτρων σε όλη την ε, Μεσόγειο Αυτό ήταν σημαντική επιτυχία, διότι ακούμε και επικρίσεις από τους αλληλείς μας στη Μεσόγειο που μας λένε ότι έχουμε άμεσο ανταγωνισμό, έχουμε συναγωνισμό με άλλους αλληλείς που δεν πρέπει να υπακούν τους ίδιους κανόνες. Πιστεύω ότι αυτή η πτυχή είναι πολύ σημαντική, πρέπει να υπογραμμιστεί και είμαστε εδώ για να απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις τεχνικής φύσεως και άλλες που θα μπορούσαν να υποβληθούν σχετικά με αυτόν τον κανονισμό. quería para... porque es que tampoco he entendido muy bien lo que ellos... Ε, δεν κατάλαβα πολύ καλά τι προτείνουν. Αν είναι αδύνατη η τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων. Άρθρο, το παλιό άρθρο 9, αν θυμάμαι καλά. Δεδομένου ότι ε, ελάχιστες Τροποποίηση έγιναν σχέση με τον παλιό κανονισμό σε ορισμένα εργαλεία που πραγματικά ήταν πολύ βλαβερά και συμφωνώ. Αλλά στο, στο διατακτικό υπάρχει δίδεται δυνατότητα παρέκκλησης προς τα κράτη-μέλη αν ε, τηρούνται ορισμένα κριτήρια. Οπότε δεν καταλαβαίνω το παράπονο Αν υπάρχουν λόγοι, βάσιμοι λόγοι, μπορεί το κρατημένο να ζητήσουν παρέκκληση. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν πολύ καλά. Εγώ ήμουν συγκίτρια σε αυτό το θέμα και συζητήσαμε πολύ κοντά, πολύ στενά με την Κομισιόν. Ε, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όταν υπάρχει επαρκής αιτιολογία, μπορεί να τροποποιηθεί ο κανόνας. Ο κανονισμός προβλέπει αρκετή ελαστικότητα. και προέχει και άλλα σημεία που προσδίδουν ελαστικότητα ο κανονισμός αυτός σε περίπτωση που επιστημονικά στοιχεία δείξουν ότι μια τεχνική είναι πολύ βραβερή κλπ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν τα πρόβλημα. Μετά, είπατε για, για, τον, 40 μιλίμετρα, ε, μιλάμε για την ρομβοειδή ή για, τη, για, για ρομβοειδές ή για το τετράγωνο μάτι. Μιλώ για τη Γενική Επιτροπή Αλίας στη Μεσόγειο. Ε, δεν είναι σαφές αυτά τα 40 μιλιμέτρα σε τι αναφέρονται, στο ρομβοειδές μάτι ή στο τετράγωνο μάτι. Δεν ξέρω τι, σε, τι αναφέρει η Γενική Επιτροπή Αλίας. Ε, Κομισιόν, έχετε δίκιο. Ε, ο οργανισμός έχει ε, ελαστικότητα. Τα κράτη-μέλη μέσω των επαφών τους με τις ε, ενώσεις αλλιέων κλπ. κατά την κατάρτιση των εθνικών προγραμμάτων διαχείρισης μπορούν να ζητήσουν τις απαραίτητες αποκλήσεις για την δική τους τοπική αλία υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για να την, τις αιτιολογήσουν επαρκώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ερώτησή σας, υιοθετήσαμε την σύσταση στην Γενική Επιτροπή Αλία ε, για τη Μεσόγειο με τους ίδιους ακριβώς όρους. τα μέλη της ε, Γενικής Επιτροπής Αλίας ε, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ή ένα τετράγωνο μάτι 40 mm ή ένα ρομβοειδές μάτι 50 mm. Τον ίδιο κανόνα δηλαδή, τον οποίο έχουμε και εμείς. Κύριε Φράγα. Αυτό με τα 3 μιλιμέτρα ε, έχει, έχει σχέση με, με συγκεκριμένα εργαλεία. Α, εγώ, ε, ναι, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ναι. Είχα κάποιες αμφιβολίες, αλλά εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ σε όλους που μείνατε μέχρι το τέλος. Στις 3 το απόγευμα ξεκινάει η ακρόαση. Ευχαριστώ.